Okay, colleagues, can I bring the... Σύντροφοι. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Και πρώτα απ' όλα, ρωτώ εάν σας ικανοποιεί το σχέδιο της τη διάταξης. Όχι. Όχι, Πρόεδρε, ο κύριο Κράμερ, διότι άλλαξε πολύ βραχυπρόθεσμα. Στην τελευταία συνεδρίαση άρχισε πίεση να ψηφιστούν τα πάντα. Και ήταν σαφέ, το είχα πει, ότι συγκεκριμένα κομμάτια πολιτικής, το είχα υπολογίσει τουλάχιστον, δεν θα ήταν έτοιμα, το Συμβούλιο ασκεί πιέσει, το Κοινοβούλιο ασκεί πιέσει, τουλάχιστον να ε, κλείσουν τα τεχνικά ζητήματα. Και ε, έχουμε υποστεί πιέσει να κλείσουμε τα θέματα αυτά σε αυτή την νομοθεσία, σε αυτή την ε, θητεία. Δεν είμαι λοιπόν έτοιμος και επιπλέον με όλη την προσπάθεια που έχω κάνει και με όλη την πίεση του χρόνου λαμβάνω μια επιστολή από τους τουριστές. Λοιπόν, εγώ παρακαλώ εδώ πέρα τώρα να γίνει ψηφοφορία για το αν αύριο τουλάχιστον θα έχουμε κλείσει, θα μπορέσουμε να κλείσουμε το τεχνικό κομμάτι. Τώρα να ληφθεί ψηφοφορία. Καλώς. Για να εξηγήσω, οι μεγάλες ε, πολιτικές ομάδες ζήτησαν την αναβολή. Ε, Ρώτησα τη γνώμη των λοιπόν ομάδων, ΕΛΚ, φιλελευθέρων που συμφώνησαν με την αναβολή. Ενημέρωσα στη συνέχεια όλους τους συναδέλφους για την πρόταση αυτή και ξέρω ότι θέλαν να αναβληθούν όχι κάποια από τα θέματα, αλλά όλα τα θέματα. Γι' αυτό και λήφθη η απόφαση, κύριε Αλκαντράουι. Πολύ σύντομα. Και η ομάδα του κύριου Κράμερ μου ζήτησε σε μένα προσωπικά την αναβολή του δικού μου θέματος. Και οι άλλες ομάδες επίσης ε, έκριναν ότι χρειάζεται ε, λίγος περισσότερος χρόνος για να κλείσουν τα θέματα. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερε ευαισθησίε ενδεχομένω, κυρίω στα πολιτικά ζητήματα, αλλά και για τα τεχνικά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να εξετάσουμε τις προτάσεις, τις συμβαστικές προτάσεις. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μία πρόταση την οποία φαίνεται να υιοθετεί η πλειονότητα των συναδέλφων. Εγώ έχω προετοιμαστεί για μία ψηφοφορία, αλλά όχι, όχι, για αύριο. Ιδάλλως θα αναγκαστούμε να καταψηφίσουμε την, ε, τις συμβαστικές προτάσεις. Πράγμα που είναι κρίμα. Με τόση δουλειά που έχει γίνει από τον εισηγητή. Προτείνω λοιπόν και ελπίζω να συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο μερικές εβδομάδες ώστε να εξετάσουμε με όλη την απαιτούμενη γαλήνη και ηρεμία τα ζητήματα, τις συμβαστικές προτάσεις και ενδεχομένω η ψηφοφορία μπορεί να γίνει το Δεκέμβριο Ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι θα προχωρήσουμε, θα προωθήσουμε λίγο πιο γρήγορα τεχνικό θέμα. Αλλά πάντως πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα για το σύνολο των προτάσεων. Ευχαριστώ. Mr. Kuhn, do you want to speak? Ο κύριος Κούν θέλει να λάβει το λόγο, εκπροσωπεί τον κύριο Γκρός. Οι πράσινοι λοιπόν ζητούν ψηφοφορία για την ημερήσια διάταξη. Αυτή είναι η κατάσταση. Εξήγησα την ε, κατάσταση. Ο κύριος Αλκαντράου είχε ζητήσει την αναβολή. Κύριε Γκρός, έχετε το λόγο. Ή αν αναβάλουμε, να τα αναβάλουμε όλα, ναι. Και αν το Δεκέμβριο έρθουμε στην ίδια κατάσταση, σας ενημερώνω αύριο ποιες θα είναι οι θέσεις του ΕΛΚΑ. Πάντως μέχρι τώρα ε, είχε τη θέση το ΕΛΚ ότι είναι καλό να μείνει το πακέτο όπως έχει, αλλά μπορεί μέχρι τον Δεκέμβριο να αλλάξουμε γνώμη στο θέμα αυτό. Πάντως, με δημοκρατικές διαδικασίες θα ληφθεί η σχετική απόφαση και θα ζητήσω τους συναδέλφους να τοποθετηθούν. Ε, καλώς. Ε, ελπίζω μέχρι τον Δεκέμβριο να, είμαστε θέση να ψηφίσουμε όλες τις εκθέσεις, λέει ο Πρόεδρος γιατί χρειάζεται να δώσουμε και τις επιπλέον αυτές τρεις εβδομάδες. Και η πρόταση του κύριου Αλκαντράουι βέβαια σε αυτό εστιάζεται. Ο κύριος Ρικέ. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις απόψεις των άλλων γιατί άκουσα και εγώ τον ε, συντονιστή αλλά ίσως ήταν ξεχωριστό το πακέτο και ξεχωριστή η άλλη αντίδραση που δεν μου φαίνεται λογική όμως η πολιτική αντίδραση ως προς την νομοθετική διάσταση του θέματος. Δεν θέλω λοιπόν να τοποθετηθώ για το αποτέλεσμα της συμβαστικής λύσης. <clears throat> Νομίζω το πιο λογικό είναι να πούμε ότι χρειάζεται χρόνος. Αλλά το να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία το βρίσκω ούτε επιθυμητό ούτε επιθυμητέο. Δεν μπορούμε να δούμε ένα μέρος της δέσμης μέτρων του πακέτου ως ε, κάτι που θα αποκλειστεί ή όλο θα το ψηφίσουμε ή τίποτα. Ευχαριστώ. Πρόθεσή μου είναι αν συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη να γίνει η ψήφιση για το συνδρομικό πακέτο στις 17 το πρωί και να δούμε και την έκθεση back για τα δικαιώματα των επιβατών το απόγευμα. Έτσι θα έχουμε ολόκληρη την ημέρα για ψηφοφορία. Αλλά σε αυτή τη φάση αυτό είναι η βασική μου πρόταση. Κύριε Κράμερ, γρήγορα. Καταρχά, έχουμε πάνω από 4.000 τροπολογίε. Εάν χωρίσουμε το πακέτο, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε φέρει και θέματα τεχνικά πολύ δύσκολα την τελευταία περίοδο, ακριβώς επειδή έλεγες εσύ, ε, Brian, ότι πρέπει να ψηφίσουμε αύριο. Λοιπόν, κάναμε πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε διαφορετικά κάνει για να μπορέσουμε να, να ψηφίσουμε. Το τεχνικό κομμάτι δεν είναι τόσο προβληματικό. Το άλλο έχει πολλές δυσκολίες. Και γι' αυτό πρέπει να τα χωρίσουμε. Και αυτό είναι και λόγο για τον οποίο ασχολούμαι. Πέντε είμαστε, πέντε είναι οι ομάδε, δεν είναι τρει. Δεν μπορούν μόνο οι τρει να τοποθετούνται και να λαμβάνουν αποφάσει. Και αυτό που βλέπω και από τις πολιτικές ομάδες δεν συμφωνούν οι πάντες. Λοιπόν, δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι δυνατόν τέτοιου είδους σοβαρές αποφάσεις να λαμβάνονται και στις 17 πάλι δεν θα είμαστε έτοιμοι. Εάν λοιπόν το Συμβούλιο στην παρούσα αθητεία ε, θέλει να ασχοληθεί μόνο με το τεχνικό κομμάτι, γιατί είναι πιθανό να μην είναι έτοιμο, έστω. Μένουν τα υπόλοιπα όπως έχουν μέχρι τώρα. Γιατί δηλαδή ε, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα 10 και να χάσουμε τα 5, αφού ε, μπορούμε να περάσουμε το τεχνικό κομμάτι χωρίς δυσκολία. Το να ε, συνδέουμε τα δύο τμήματα της εκθέσεως για λόγους μόνο δογματικούς, θα μας οδηγήσει στην καταστροφή στο θέμα αυτό και τελικά σε πολύ μεγάλα προβλήματα πίεσης. Έχουμε και τις εκλογές ε, στο προσκήνιο και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε όχι για το περιεχόμενο, για τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Για τις 17 του μηνός τους ή άλλως πάλι θα μπορέσουμε να λάβουμε απόφαση, πάλι θα ασκήσει πιέση στο Συμβούλιο και πάλι θα μπορέσουμε να κλείσουμε το τεχνικό θέμα. Ο κύριος Φαντάλεν ήθελε το λόγο πιστεύω και αυτός. κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι πολλοί αυτοί που είχαν αντιρρήσει σε σχέση με αυτό το σημείο στην ημερήσια διαταξή, οπότε καταλαβαίνω την έτσι του, το αίτημα του κ. Κράμερ για την ψηφοφορία και σε σχέση με αυτή την αλλαγή προ την έγκριση της ημερήσιας διαταξής. Την πρόταση αυτή, την πρόταση για την ημερήσια διαταξή την λάβαμε ήδη και θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω με τον κ. Κράμερ. Κύριε Φεντάλεν, δεν υπήρξε ούτε ποτέ αμφιβολία για το ότι αν ζητά μια ομάδα ψηφοφορία την κάνουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Η ψηφοφορία προβλέπεται. Απλώ να εξηγήσω τι έλεγα. Την περασμένη εβδομάδα μου ζητήθηκε από μια ομάδα να αναβληθεί η ψηφοφορία για το συνδρομικό πακέτο. Ολόκληρο το πακέτο. Και μετά Μίλησα με το ΕΛΚ, μάλλον οι σοσιαλιστές και δημοκράτες ρώτησαν το ΕΛΚ και οι φιλελεύθεροι συμφώνησαν με την αναβολή. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι εάν οι τρεις βασικές ομάδες ζητούν αναβολή, πρέπει να ενημερώσουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό κάνω. Έτσι κι αλλιώς, και το ένα να κάνω και το άλλο, πάλι με μένα θα τα βάλετε. Οπότε μου φαίνεται Τρελό να περιμένουμε ως σήμερα. Και να μην ενημερωθούν οι άνθρωποι που έρχονται από τέτοιες μεγάλες ε, διαδρομές και ταξίδια για να ακούσουν ότι τελικά υπάρχει αναβολή ενώ θέλανε να γίνει ψηφοφορία. Έτοιμα λοιπόν του κυρίου Κράμερ να μην εγκριθεί η σε διάταξη. Οπότε το πρώτο για το οποίο θα πρέπει να ψηφίσουμε ή όχι είναι το αν θα συμφωνήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Εάν συμφωνείτε να αναβληθεί η ψηφοφορία, θα εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Εάν διαφωνείτε, θα ψηφίσετε όχι. Όπως ο κύριος Κράμερ δηλαδή. <clears throat> Εντάξει. Είναι σαφές για όλους. Όσοι είναι υπέρ της έγκρισης του σχεδίου ημερησίας διάταξης όπως έχει τυπωθεί, παρακαλώ. Κατά. 10 προς 4 υπέρ της ε, ημερήσιας διάταξης. Να προχωρήσω λοιπόν τώρα. Εάν συμβείτε ακριβώς το ίδιο 17 του μηνός την επόμενη φορά, τότε αναβάλλονται τα πάντα, έτσι δεν είναι. Ή αλλιώς μπορούμε να αποφασίσουμε στις 17 ότι θα κοιτάξουμε το τεχνικό κομμάτι μόνο. Όχι, θέλω να το ξέρω από τώρα, εάν είναι έτσι. Νομίζω, σωστό θα ήταν να πούμε, Μάικλ, ότι θα γίνει στις 17 η πλήρης ψηφοφορία για όλο το πακέτο. Εάν όχι, εγώ ως πρόεδρος θα εμείνω να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία για τις εκθέσεις που είναι έτοιμες μόνον. Δεν μπορούμε να χασομεράμε. Έχεις απόλυτο δίκιο όταν λες ότι πίεζα για να είμαστε έτοιμοι για σήμερα ή αύριο. Δίκιο έχεις, έτσι είναι. Αλλά δεν ήταν για προσωπικούς λόγους. Δεν ζήτησα εγώ την αναβολή. Βάσει όσων λέει για το ΕΛΚ και ο κύριος Γκρός και για το τι άποψη μπορεί να έχουν στις 17, δεν είμαι και ικανός να διαβάζω κρυστάλλινες σφαίρες, δεν είμαι μάγος και να ξέρω τι θα αποφασίσουν, αλλά είναι σαφές ε, με όλους τους συντονιστές με τους οποίους μίλησα και μου έβαλαν ε, το αίτημά τους, είναι σαφές για όλους. Πρέπει να ψηφιστεί αυτό στις 17 Δεκεμβρίου. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Εντάξει. Ωραία. Έγκριση πρακτικών. Σας αρέσουν τα πρακτικά σε όλους. Ωραία. Τώρα, αν ανακοίνωση του Συμβουλίου για τον ταχόγραφο. Η θέση του Συμβουλίου ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια στις 21 Σεπτεμβρίου 2013, κανόνας 163, ε, άρθρο 163 του καταστατικού. Η θέση του Συμβουλίου θα περιληφθεί ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης της αρμόδιας επιτροπής μετά, ε, στη συνεδρίασή της μετά την ημερομηνία αυτή. το σχέδιο σύστασης της κυρίας Τσικάου για δεύτερη ανάγνωση θα συζητηθεί αύριο το απόγευμα. Και να σα θυμίσω ότι το κείμενο που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο αντικατοπτρίζει τη συμφωνία που επετέφθη μεταξύ των εισηγητών, των σκιωδών και του Συμβουλίου. Ενημερώνω του συναδελφού ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι την 5η στι 28 Νοεμβρίου στι 12 το μεσημέρι, προκειμένου να μπορέσει η ψηφοφορία να γίνει στι 17 Δεκεμβρίου, μία ημέρα αφιερωμένη στι ψηφοφορίε και να περάσει στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο. Έπρεπε να γίνει και αυτή η επίσημη ανακοίνωση. Επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψεων με τους συντονιστές των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ξεκινάμε με τους πρώτους πέντε σήμερα το απόγευμα. Να με, συγχωρήσουν οι συντονιστέ αν, αν κάποια στιγμή χρειαστεί να φύγω. Ε, πρέπει να πάω και σε άλλα σημεία του Κοινοβουλίου σήμερα. Αλλά θα με αντικαταστήσει ο Αντιπρόεδρο. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε τι αιτήσει εκθέσει των συντονιστών σήμερα για τα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Πρώτος ο συντονιστής ο κύριος Κόξ για το Priority Project, το σχέδιο προτεραιότητας παριθμών 1. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξέτομα βουλευτές, χαίρομαι που μπορώ να είμαι σήμερα εδώ. Ολοκληρώνεται η πρώτη μου εντολή ως ε, συντονιστή. Ξεκίνησε το 2010, παρατάθηκε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του τρέχοντος. Τεχνικά λύγει και το πρώτο πρόγραμμα προτεραιότητας που με βάση και τις κατευθύνσεις γραμμές και το μέσο Connecting Europe θα είναι ο πέμπτος διάδρομος, σκανδιναβικός μεσογειακός διάδρομος στο βασικό δίκτυο. Θέλω να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι ήθελα να επικεντρωθώ στα οικονομικά. Να σας πω ότι σημειώσαμε πρόοδο. 18 Απριλίου του 2011 σας υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα με τη σύραγγα του Μπρένερο συγκεκριμένα έφτασε ε, σε ένα διέξοδο. Έπρεπε το BBTSC, η εταιρεία δηλαδή που είχε αναλάβει την ανέγεση της σύραγγας, ε, ε, να συμφωνήσουμε για την ανακατανομή, αναδιαμάλων του κόσμου μεταξύ ιδίως Αυστρίας και Ιταλίας. Η Αυστρία δεσμεύτηκε να δώσει πάνω από 1,5 δις από το 2013-2018 για το BBTSC 635 εκατομμύρια από την Ιταλία για τα επόμενα δύο χρόνια, 297 μέχρι το τέλος 2017 και έχουμε και 338 για τον αυτοκινητόδρομο Α8. Υπάρχουν βέβαια κάποιες διαφορές στην Ιταλία ε, και δεν έχει προχωρήσει η εκταμίευση αυτών των πόρων, πάντως θα δετεθούν τα χρήματα αυτά. Να πω κάτι ακόμη για τα οικονομικά. Δυστυχώς όπως γνωρίζετε σε ορισμένα κράτη-μέλη και η Αυστρία περιλαμβάνεται και μάλλον και η Ιταλία, συνεχίζεται η πολιτική λιτότητα, οπότε δυνητικά μπορεί κανεί να αναμένει περαιτέρω ανάγκη περικοπή των δημόσιων δαπανών που μπορεί ή, να, και μπορεί να μην, αλλά ενδεχομένω και να επηρεάσει ε, την πρικοδότηση αυτού του project ε, και το κατά πόσο θα είναι έτοιμο έγκαιρα. Πού βρίσκεται τώρα ε, η πρόσφαση των εργασιών. Περιμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί εργασίε τη έργα του Μπρένερο να έχουμε 200 για χιλιόμετρα. Έχουμε ένα προ, ε, μία σύραγγα πρόσβασης και άλλα έργα, 14% έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή 28 χιλιόμετρα και των οποίων δύο, των δύο βασικών σειράγγων στο Ιταλικό τμήμα. Στη γραμμή μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, στο περιαντριατικό ρήγμα. Τα πράγματα πάνε καλά, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες. Ε, η Ιταλία και η Αυστρία έχουν κάνει ό,τι μπορούν σε αυτή την περίοδο της λιτότητας και το Εποπτικό Συμβούλιο της BBTC τον Ιούλιο δεσμεύτηκε να ξεκινήσουν τρεις ακόμη παρτίδες. Έχουμε τρεις προκέξεις διαγωνισμών, ε, ένα δις ευρώ. Άρα έχουμε σημαντική πρόοδο να σας αναφέρουμε. Τώρα, τι γίνεται με τι βόρειες και νότιες οδεύσεις. Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, είναι το πιο δύσκολο, αυτή η παρτίδα <clears throat> νοτίως του Μπρένερο, νοτίτσα μέχρι Πόντε Καρντένα. Είχαμε την πρώτη φάση σχεδιασμού και περνάμε στην ύστερη φάση σχεδιασμού τώρα. Έχουμε σημαντική πρόοδο και μάλλον ε, το 2016-2017 θα ξεκινήσουν ε, οι εργασίες. Βέβαια δεν θα ολοκληρωθεί, δεν θα παραδοθεί αυτό το σημείο πρόσβασης σε έγκαιρα. Τώρα σε ό,τι αφορά τη βόρεια ε, διαδρομή, το Δεκέμβριο πέρυσι 34 χιλιόμετρα άνοιξαν στην Αυστρία. Πολύ σημαντική αυστριακή λοιπόν συμβολή ε, για την οδό αυτή. Αυτό το οποίο παραμένει τώρα είναι το νοτίος ε, του Μονάχου στο Κίφερ Στέλντεν τμήμα όπου τον Ιούνιο πέρυσι εκεί είχαμε μια διπουργική απόφαση μεταξύ του Υπουργού Ραμσάρ και του Υπουργού Μπίρεσιφ, ε, Γερμανού και Αυστριακού, για τον πρόωρο σχεδιασμό που έπρεπε να ξεκινήσει, για τη μελέτη, την προμελέτη που έπρεπε να ξεκινήσει 3,4 δις παρέχουμε ε, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ε, για αυτό το διαγωνισμό, στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεν έχει όμως γίνει ακόμη το έργο αυτό και περιμένω τη 10η Δεκεμβρίου γιατί θα συναντηθώ τότε με τον νέο Υπουργό ε, της Βαβαρίας για τις μεταφορές, ε, τον κύριο Χέρμαν. Και όταν θα έχουμε και νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο, την Ομοσπονδιακή, ελπίζω να συναντηθώ με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών στο Βερολίνο. Να έρθω τώρα στα συνοδευτικά μέτρα, δηλαδή τι κάνουμε για να αναπτύξουμε τη δομή της πολιτικής. Φόροι κατανάλωσης, διόδια, ε, τι κάνουμε για να τα αναπτύξουμε εκ παραλλήλου με τις νέες υποδομές. Νομίζω ότι η πολιτική μηχανική με ήττα θα είναι ίσως και πιο δύσκολη από, την, ε, από τα έργα πολιτικού μηχανικού. Στις 25 του Σεπτεμβρίου φέτος το πρωτόκολλο μεταφόρων της ε, Σύμβασης των Άλπαιων τέθηκε σε ισχύ Πρόκειται για μια πρωτοβουλία δική μου ε, σε συνδυασμό και με την Ιταλική κυβέρνηση όταν έφυγε από την κυβέρνηση το κόμμα του Μπόση. Πέρασε λοιπόν πέσει στην Ιταλία. Το πρώτο ήμιση αυτού της χρονιάς κινητοποιήθηκε και η Ιρλανδική Προεδρία για να επικυρώσει Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, και τώρα πλέον έχει τεθεί σε ισχύ αυτό που σημαίνει ότι πλέον έχουν όλοι τις ίδιες αρχές, για τη σύμβαση των Άλπαιων δηλαδή, σε ό,τι αφορά και τα συνοδευτικά μέτρα. Δεν θέλω να υπερεκτιμήσω ε, τις επιπτώσεις, αλλά σε διάφορου τομεί πολιτική ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όλοι να ε, ακολουθήσουν τις ίδιες γραμμές ε, από όλε τις περιφέρειες, από όλες ε, τις περιοχές. Κύριε Πρόεδρε, να περάσω σε κάτι άλλο. Ο νέος διάδρομος ε, θα έχει ένα σημείο ε, συμφόρησης ε, που θα είναι η διασύνδεση μεταξύ Δανίας και Γερμανίας. Αυτό θα έρθει μαζί με τη σύραγγα του Μπρένερο. Είναι τα σημαντικότερα στοιχεία του πέμπτου διαδρόμου του βασικού δικτύου. Για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης θα έχουμε συντονιστές θα έχουμε μια μελέτη χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πρόγραμμα εργασίας που θα ανακύψει και θα υπάρξουν και πολλές συνδριάσεις του φόρουμ για το μετοδιάδρομο. Τώρα σε ό,τι αφορά το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη, το Connecting Europe, ε, έχουμε 11,2 δις από τα 26 δις ήδη ε, στα κράτη συνοχής, μένουν 14,8 δις είναι σημαντικό το ποσό, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την κλίμακα των φιλοδοξιών που έχουμε στο σχεδιασμό των μεταφορών, δεν είναι και τόσο μεγάλο τελικά αυτό το νούμερο, γιατί πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μα πόσα κράτη ενέχονται, πόσοι τρόποι μεταφορών και πόσα χρόνια. Άρα πρέπει να βρούμε καινοτόμο χρηματοδότηση εκτό των χρημάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να μοχλευθούν ε, επιτάνω προς τα άνω. Τώρα, σε ό,τι αφορά πάλι την πολιτική, έρχομαι στο θέμα της επικοινωνίας. Κάθε χρόνο, σας το τονίζω αγαπητέ Πρόεδρε, κάνουμε φανταστική δουλειά, γεωλογικές μελέτες, ε, υδρογεωλογικές μελέτες, μελέτες ε, πολιτικού μηχανικού, βελτιστοποίηση, χρηματοδοτικά ε, προγράμματα κτλ. κτλ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τελευταίο για την επικοινωνία. Το είχα πει και με το, το συνδρομικό σταθμό της Ουτγάρδης ε, στη Γερμανία. Όταν ε, έπρεπε να παραδοθεί το έργο αυτό, είχαν κουραστεί όλοι πλέον, υπήρχε κόποση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική επικοινωνία, ε, ώστε η μητρότητα, η πατρότητα να είναι κάτι γενικό και να μην συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και την Επιτροπή σας ε, για την ε, προσωπική σας δέσμευση ε, και τη συνεργασία που είχαμε και προσωπικά. Και τον Λίγο Χούμπερτς από την ΓΔΜ της Κομισιόν θέλω να τον ευχαριστήσω και να πω σε όσους σε όσους ε, θα ε, συμμετάσχετε στις επόμενες εκλογές κάθε επιτυχία και σε όσους δεν συμμετάσχετε πάλι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόξ. Έχουμε δώσει 25 λεπτά για το καθιστούνιστε. Κύριε Λίχτον Πέργερο, κύριος Κράμερ, έτερος. Για να κάνει ερωτήσεις, καν του συνάδελφοι. ερωτήσει όμως είναι δυνατόν, όχι ομιλίες. Κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόξ. όντω πολύ διεξοδική η έκθεσή σας, πολύ μου άρεσε. Και ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναφέρεστε στην ε, διαδρομή πρόσβασης. Έχουμε το Σεν Κοτάρ σχεδόν έτοιμο τώρα. Αλλά για πρόσβαση δεν ακούμε τίποτα ούτε από την Ιταλία ούτε από τη Γερμανία. Ούτε κουβεντούρα λοιπόν όπως λέμε και στην Αυστρία ε, και όμως χρειάζεται να γίνουν οι δρόμοι πρόσβασης. Ιδάλλως έχουμε να κάνουμε με μία με έναν καθεδρικό στην έρημο, όπω λέμε στο Νότιο Τυρόλο, ότι δηλαδή έχουμε φτιάξει ένα μεγάλο έργο χωρί όμω να εξυπηρετεί το βασικό στόχο για τον οποίο έχει οικοδομηθεί. Και γι' αυτό παρακαλώ, ιδιαίτερα για τι προσβάσει να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια με τη στράτευση που σας χαρακτηρίζει. Αναφερθήκατε λοιπόν στις προσφάσεις σε σχέση με τη Γερμανία. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας όντως μεταξύ των δύο Υπουργείων, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποιο συμμετέχει. Πρόκειται για το Ομοσπονδιακό ε, Υπουργείο των Μεταφορών. Είναι τα περιφερειακά δηλαδή των κρατηδίων που εμπλέκονται στις διαδρομές αυτές. Πού, που, που έγκυται η σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί τη Βαβαρία και το Νότιο Τυρόλο όπως και το Τρεντίνο τα, τα γνωρίζω αρκετά καλά και θα ήθελα να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διότι είμαι πάρα πολύ βεβαία ότι ε, θα χρειαστεί σοβαρό σχεδιασμό για τι διαδρομέ πρόσβαση. Λέτε στην έκθεση ότι από την πλευρά τη Ιταλία οι Ιταλικοί σιδηρόδρομοι επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του. Confirms its intention. Να κάνουν το εξή κτλ. Ναι, ε, όμω να σα πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει τίποτα ή ότι πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Περιμένω να κάτι από το. Και με ιδιαίτερη ε, εκτίμηση σημειώνω ότι έχετε εντοπίσει τα διάφορα στάδια της υλοποίηση και πρέπει να τα, παρα, ε, να, τα, να τα καταμετρήσουμε, να τα παρακολουθήσουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι τελικά θα γίνει κάτι στην ουσία γιατί η Ιταλία είναι ακόμα στην φάση πριν το σχεδιασμό, είναι στα προσχέδια και μπορεί να κρατήσουν δεκαετίες ακόμη τα έργα αυτά πριν να υλοποιηθούν. Κάτι ακόμη το οποίο αναφέρατε και το οποίο θεωρώ εξίσου σημαντικό όπως και εσείς και το πρόβλημα το πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι το εξής και αποδεικνύεται ότι Μπορεί να υπάρχει η Βερόνα στην Ιταλία, αλλά δεν τρέχουν όλοι συλλήβδινοι επιβάτες να, να, να, φτάσουν στη Βερόνα, αλλά περνάνε από την Ιταλία από την άλλη μεριά οι μεγάλοι άξονες. Και έχουμε ακόμη ανάγκη να φτιάξουμε ε, διαδρομές για μεταφορά φορτίων. Πολλές ακόμη υποδομές μένουν να γίνουν. Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι μπορούμε να έχουμε μικτής χρήσεως σύραγγα ή θα είναι αποκλειστικά και πάλι και μόνο σύραγγα για μεταφορά επιβατών όπως είχε αρχικά δοθεί η υπόσχεση στο Τυρόλο. Γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία, αλλά φαίνεται ότι δεν θα τηρηθεί η υπόσχεση και έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Ρωτώ λοιπόν, πρόκειται να δοθεί άδεια για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της ε, σύραγγας αυτής, εφόσον εγκαταλείψει τελείω τα φορτηγά αυτοκίνητα. Ε, και επίσης ξέρετε ότι υπάρχει διατυπωμένη επιφύλαξη σε σχέση με τη Σύμβαση των Άλπαιων για την ε, κατασκευή των έργων υποδομής εφόσον πρόκειται αυτά να ε, μεταφέρουν και εμπορεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να συντομεύσουμε λίγο τις παρεμβάσεις. Καταλαβαίνω ότι το θέμα σας αφορά ιδιαιτέρως, αλλά δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες οι δικές σας παρεμβάσεις από ότι το ίδιο του συντονιστή. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστούμε στα δύο λεπτά. Βρίσκονται αρκετό. Κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να πω ότι έχουμε μια, ένα ιστορικό δεκαετιών πίσω μας και πρέπει να σας πω για ε, Ρότερταμ Γένοβα είναι μια διαδρομή για την οποία έχει δεσμευθεί η Γερμανία από το 1996 να ε, κατασκευάσει το δικό της μερίδιο της διαδρομής και χρειάζονται ακόμα 4 δισεκατομμύρια το οποίο σημαίνει περίπου 200 χρόνια μέχρι να κλείσει η διαδρομή ε, Ρότερνταμ, ε, Γένοβα ε, και μας λέτε ότι η Γερμανία διαθέτει πολλά λεφτά. Πολύ καλά, αλλά υπάρχουν κάποιες αναφορές στο γερμανικό τύπο ότι χρειάζεται μετά από μια επιθεώρηση να ανακαινιστούν 1.400 γέφυρες το χρόνο, πράγμα το οποίο σημαίνει με, μια, με ένα αριθμό περίπου 100 ε, το χρόνο ότι χρειαζόμαστε περίπου 12-12 χρόνια για να κλείσει όλη αυτή η υπόθεση. Και μετά μην ξεχνάμε τις υπόλοιπες διαδρομές και τα σημεία στα οποία έχουμε την, ε, έχουμε την ανάγκη να υποταχθούμε βεβαίως και στις επιταγές του ε, οικοδομικού δικαίου και που πρέπει να τηρήσουμε κάποιες διατάξεις. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν όπως μας λέτε να ε, τιμηθούν οι 14 διαφορετικές συμβάσεις που έχει συνυπογράψει η Γερμανία και δεν μιλάω για Βουλγαρίες και Ρουμανίες, μιλάω για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας η οποία υποτίθεται ότι έχει λεφτά ε, και όμως δεν μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει να λάβει μέσω της, ε, των συμβάσεων αυτών. θα τα καταλήξουμε δηλαδή με ένα συνονθήλευμα από, από κομμάτια σιδηροδρομικού δικτύου ε, από κομμάτια ε, οδικών μεταφορών ένα, μια κουρελού ουσιαστικά, ένα μοσαϊκό το οποίο θα αποτελεί δίκτυο ε, δίκτυο μεταχωρών. Και θα ήθελα να αναφέρω και το παράδειγμα εκείνης της, εκείνου του κομματιού του δρόμου που έκανε 25 χρόνια για να ανασκευάσει η Γερμανία για 600 ακριβώς 600 ε, μέτρα, 660 μέτρα που χρειάστηκαν να γιατί είχαν καταστραφεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πέρασαν 25 χρόνια για να υλοποιηθεί η ανασκευή. Το ίδιο με τη γέφυρα Φιμάλβερ με το Ρόστοκ όπου υπάρχει κόμβος πρέπει να αξιοποιηθεί ο, ο, ο κόμβος για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί το Αμβούργο ε, και ως εκ τούτου και οι χώρες της Σκανδιναβικής ε, Χέρσονήσου, αλλά τα 40 χιλιόμετρα που αντιστοιχούν στην ε, Δανία δεν τα υλοποιεί, δεν τα ανακαινίζει η Γερμανία για να ασκήσει πιέσεις, για να έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τη γέφυρα Φέρμαν. Έτσι λοιπόν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Οι υποδομέ βεβαίω χρειάζονται χρήματα. Ναι, πρόεδρε, σας άκουσα χρειάζεται, χρειάζεται να, να εισπραχθούν τα χρήματα αυτά, να βρεθούν τα χρήματα αυτά, αλλά πώς από τα διόδια ε, για τις ε, μεταφορές φορτίων, για τις μεταφορές εμπορευμάτων στη Γερμανία από αλλοδαπές εταιρείε. Δεν υπάρχει ένας λόγος η Γερμανία να ρίξει άλλα λεφτά δικά της, ε, ούτε καν θέλει να διευρύνει τα, τα διόδια αυτά. 60.000 πιο πολύ είναι η ζημιά, 60.000 φορές πιο μεγάλη είναι η ζημιά προξενή στο οδικό δίκτυο ένα φορτηγό αυτοκίνητο από ότι ένα ιδιωτικής χρήσης, ένα μικρό επιβατικό αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η συμβολή αυτών των διοδίων για τα φορτηγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Σκαντσιάν. Μια διαφορετική άποψη από τους δύο προηγούμενους συναδέλφους. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Μπατ Κόξ, ο οποίος έχει κάνει τεράστιο έργο κατά την άποψή μου, με πραγματικά φοβερή αφοσίωση, εξαιρετική. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος, αυτό, αυτό το πέρασμα από το βορρά προς τον νότο, ε, Πρέπει να παραμείνει, να πάρει σάρκα και οστά, να μην μείνει ένας πύργος στην έρημο. Διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα έχει νόημα το έργο μας. Πιστεύω ότι από το 30 διαδρόμους περάσαμε σε 9. Κάναμε προσπάθεια απλούστευσης. Έγινε πολλή δουλειά. Και νομίζω ότι καλώς έγινε και με καλό τρόπο. Όμως είναι δύο οι πτυχές που μας ενδιαφέρουν, ο σχεδιασμός και οι επενδύσεις. Ό,τι αφορά το σχεδιασμό, νομίζω ότι η κατεύθυνση που ακολουθείται είναι σωστή και πρέπει να επιταχύνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση σε σχέση με τις διάφορες τοπικές αντιφάσεις. Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, ξέρω ότι Το συζητάμε εδώ και μήνες. Είναι πολύ λίγοι οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Και δεν είναι σίγουρο ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε προγραμματίσει. Εάν όμως θέλουμε να βρούμε ε, χρηματοδοτήσεις εναλλακτικέ ή το εάν η Ευρώπη θα μπορούσε να έχει ομόλογα στο χρηματοπιστωτικό κόσμο και στις αγορές, θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και διαφορετική στάση προς τον προγραμματισμό μας και να έχουμε ελπίδες ότι περισσότερα θα υλοποιηθούν. Και τώρα για την πλατφόρμα των διαδρομών, κάτι διαφορετικό από όσο τώρα. Ακούσαμε την άποψή σας κύριε Κόξ. Αλλά πώς επιπλέον θεωρείτε ότι έχει γίνει αυτό το έργο με καλό τρόπο, θα έχουμε τις δυνατότητες και την, ε, το εργατικό δυναμικό ώστε ε, στην πράξη να υλοποιηθούν όσα με τόση δυσκολία δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε εμεί να συντονίσουμε αυτή την εργασία και να έχουμε επιπλέον κάποια δυνατότητα να φτάσουμε σε τοπικές συμφωνίες. Ήθελα την άποψή σας σχετικά. Ευχαριστούμε κύριε Καντσάν. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Έρτουκ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κόξ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση σας. Έχω μια ερώτηση ε, για τα έγγραφα από τα οποία βλέπω και είναι πολύ σημαντικό πιστεύω, ίσως λιγότερο για κάποιους άλλους, αλλά πάντως για μένα πολύ σημαντικό σε σχέση με την περαιτέρω μεθοδολογία. Λέτε στις 15 Ιανουαρίου του 2013 έλαβε χώρα μια ενημερωτική εκδήλωση για τα δίκτυα ΤΕΜΠΕ και για τις υποδομές ΤΕΜΠΕ. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αυτές οι εκδηλώσεις ενημέρωσης. Τι είδους υπόλοιποχής έτυχαν. Και δεύτερον, έγινε, ελήφθη κάποια δεσμευτική απόφαση, συμφωνία, εάν βέβαια προέκυψε συμφωνία, και εν τέλει τι είδους αποτελέσματα βλέπουμε σε σχέση με τους διαφόρους εμπλεκομένους, για τους διαφόρους εμπλεκομένους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ερτούγκ. Να δώσω το λόγο στο συντονιστή μα, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη ανταταπτοκαθυστέρηση, οπότε καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να αυτοπιθαχηθούμε. Ιδάλω. θα τσακωθούμε να έρθει πίσω ο Πρόεδρος και μα βρει έτσι. Κύριε Κόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λιχτεμπέργκερ, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το σχέδιο προτεραιότητα 1, γιατί γι' αυτό σα μιλώ σήμερα, δεν θα είναι σίγουρα πύργο στην έρημο ή τουλάχιστον αυτό δεν είναι ο στόχο. Μα Γι' αυτό σχεδιάζουμε αυτού του δρόμου πρόσβαση κτλ. Επίση, σε ό,τι αφορά αυτό και, αυτή και άλλη, άλλη σύγκριση και θα έρθω λίγο στην ε, διαλπική περιοχή εν γέννη όχι μόνο διάδρομο προς διάδρομο πρέπει γενικά να βελτιστοποιήσουμε την αυτή υποδομή είτε είναι στην Ελβετία είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος μας είναι να γίνεται corridor shopping, ε, επιλογή διαδρόμων για λάθος λόγους. Και αυτό το βλέπουμε, αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι χαμηλότερη η δική φορά κατανάλωση σε κάποια χώρα αντί για κάποια άλλη, ακόμη και αν μεταφέρεται ο θόρυβος, η ρήπανση και η κυκλοφορία σε ε, άλλες περιοχές και παραβιάζονται οι κανόνες της Ένωσης. Είναι μια πολυεπίπεδη ανάλυση αυτό που πρέπει να γίνει, αλλά συμφωνώ ότι πρέπει, πρέπει να το προσέξουμε. Σε ό,τι αφορά Και αυτό και το ερώτημα του κύριου Έρτουγκ, νομίζω. Σε ό,τι αφορά το Μόναχο, Μόναχο Αυστρία, Κίφερσφελτ, ενημέρωση λοιπά, Πράγματι, έγινε μια προκαταρτική ενημερωτική συνεδρία. Είναι όμως πάρα πολύ πρόημο. Γι' αυτό και το μόνο που θέλαμε να κάνουμε ήταν να δώσουμε ένα σήμα, αν θέλετε, ότι είμαστε ανοιχτοί να επικοινωνήσουμε αυτόν τον κόσμο και νομίζω ότι είναι και ένα σημαντικό μήνυμα ότι ε, είμαστε προσιλωμένοι στο να συμμετέχει η τοπική κοινωνία, να τους ε, δίνουμε απαντήσεις, να ακούμε τα ερωτήματά τους. Αλλά σε ό,τι αφορά τα σχέδια ευθυγράμμισης, ε, αυτή η επικοινωνία μπορεί να παραμείνει στο θεωρητικό επίπεδο γιατί κάποιος θέλει να μάθει. Περνάει από, το, ε, από την πόλη του, από το χωριό του ο δρόμος ή όχι. Πάει, ε, βυθίζεται κάπου ή παραμένει μόνο επίγειος κτλ. Ε, το να γίνει σε βάθος συζήτηση με αυτές τις τοπικές κοινωνίες είναι χρήσιμο, το λέω με κάθε ειλικρίνη, αλλά είναι πρόημο, πρόωρο κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και χρειάζονται μελέτες τις οποίες προανέφερε για τα 3,4 της, ε, της συγχρηματοδότησης ευρωπαϊκής για να δούμε αυτό το θέμα της ευθυγράμμισης ε, και της χαρτογράφησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να χαρτογραφήσουμε τις οδούς ευθυγράμμισης. Η κυρία Λίχτεμπέργκερ ρώτησε για την Ιταλική δέσμευση, ποια είναι η πρόθεση κτλ. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Ιταλικός νόμος ε, για την ευστάθεια, στα μπιλιτά, και επειδή έχουμε αυτή την ε, πολιτική λιτότητα, υπάρχει ειδική χρηματοδότηση σε αυτό το νόμο, λέτε, τη σταμπιλιτά, για το συγκεκριμένο project. Δεύτερον, με βάση το ταλικό σύστημα, για κάτι που είναι στο δημοσιονομικό νόμο πρέπει να περάσουν άλλες δύο δοκιμασίες. Υπουργική έγκριση στην Επιτροπή Τσίπε και μετά να, πρέπει, να, ελεγχθεί, και να εγκριθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Έγιναν και τα τρία αυτά. Πέρασε το, τη δοκιμή στάθειας, ε, πέρασε από την Επιτροπή ε, για τις δαπάνες και πέρασε και το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας είναι δέσμευση αυτή και είναι ουσιαστική και απτή. Και κάτι άλλο που δεν έχει κάνει κάποιο κράτος ακόμη είναι ότι έχουν ορίσει ε, τον δικό τους συντονιστή, τον κύριο Φαμπρίς. Υπάρχει λοιπόν ένας εσωτερικός συντονιστής. Αυτό αποτελεί προσθέμενη αξία. Εγώ μπορώ να γνωρίζω το Τσίπε και το ελληνικό συνέδριο, αλλά όπως ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που είναι Ιταλός δεν τα γνωρίζω. Έχουμε λοιπόν εσωτερική ενημέρωση και αυτό πραγματικά κινητοποίηση, ήταν ένας μοχλός κινητοποίησης. Σε ό,τι αφορά τα φορτία, φυσικά και στόχο μα είναι να αντιμετωπίσουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων, των φορτίων. Αν δείτε σε αυτό το έγγραφο για του διαδρόμου του βασικού δικτύου, θα δείτε ότι για το διάδρομο 5 τα πάντα σχεδόν είναι λιμάνια σιδηρόδρομοι, οι λεγόμενοι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι Αυτά τα τρία είναι για το μέλλον και όχι οι οδικές αρτήριες τόσο. Βέβαια υπάρχουν και ζητήματα διατροπικότητας και γιατί σας το τονίζω αυτό. Γιατί αυτή είναι, ε, αυτό είναι το επίκεντρο, αυτή είναι η εστίαση που έχουμε και αυτή είναι η εντολή μας για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Για τη Βερόνα, ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο διασταύρωσης, διασταύρωσης ε, βορράς νότου, νότος, ε, δύση, ανατολή. Αλλά πράγματι είναι πολύ σημαντική η Βερόνα. Τώρα εσείς ίσως στην επιτροπή σας δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Quadrante Europa που είναι μια τεράστια εγκατάσταση ε, χειρισμού ε, φορτίων. Εγώ έχω δει ότι μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου και των συνδρομικών εταιριών έχουμε πολύ διαφορετικές ε, στάσεις, συμπεριφορές και ενώ λένε όλοι ότι είναι ανοιχτή προς όλους, είναι ανοιχτή μόνο λίγες ώρες της μέρας της νύχτας. Και δεν έχουμε αυτό το βαθμό της φιλελευθεροποίησης με την έννοια ότι δεν υπάρχει ε, επαρκές άνοιγμα ε, όλων προς όλους. Άρα έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα. Για τον κύριο Κράμερ μιλήσατε για πολλά πράγματα, τον αριθμό των ε, διαδρόμων, είσοδος έξω από τη Γερμανία, ρετροφίτ κτλ. Η Γερμανία είναι στο ευρωπαϊκό κομμάτι και έχει, κάνει τεράστιες, ε, έχει αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις. Πρέπει να σας πω ότι στο Διεθνό Φόρο Μεταφορών στη λυψία. ο Υπουργείο Ράμσο είχε επιβεβαιώσει σε σχετικό ερώτημα ότι η βασική πρόκληση για τη Γερμανία την επόμενη δεκαετία είναι η συντήρηση και η ανανέωση της υφιστάμενης υποδομής και όχι ε, η πρόθεση νέων projects. Άρα πράγματι εκεί υπάρχει ένα θέμα ότι δεν είναι προτεραιότητά τους ε, και θα έχουμε διαπραγματεύσεις με τη γερμανική πλευρά, δεν θα είναι εύκολες. Ε, θα δούμε ποιες είναι οι δεσμεύσεις. Βέβαια έχει προσυπογράψει η Γερμανία, άρα έχει δεσμευτεί. Αλλά για τις γέφυρες που είπατε, δεν είναι μόνο οι γέφυρες και άλλες υποδομές, το επίπεδο τη χρηματοδότηση ε, ω ποσοστό του ΕΠ που απαιτείται μόνο για τη συντήρηση και την ε, ε, επισκευή επιδιόρθωση είναι τεράστιο. Έγιναν βέβαια πάρα πολλά όταν ήταν η εποχή του οικονομικού θαύματος της Γερμανίας, αλλά έχουν παλιώσει οι υποδομές. Επίσης και για το νότιο του Μονάχου και για κάποιο άλλο κομμάτι που ρωτήσατε, η ευθυγράμμιση, η χάραξη είναι σαφής, ε, μπορεί να τα δει αυτή, αυτά κανείς στους χάρτες. Υπάρχει σίγουρα ε, στο TBNet, ε, στο δίκτυο της Deutsche Bank, η σκέψη αν κάποιες διαδρομές φορτίων αποχωριστούν για ένα κομμάτι και μετά ξαναμπούν στη γραμμή υψηλής δυναμικότητας. Εγώ Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το αν θα γίνει όχι, αλλά ξέρω ότι το σκέφτονται. Ο κύριος Καντσιάν ρώτησε για τους διαδρόμους και αν είναι εφικτό. Αν διαβάσετε κύριε Κάντσιαν αυτό το έγγραφο για το πέμπτο διάδρομο, η έφαση δίνεται στους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους, στα λιμάνια και στους σιδηρόδρομους. Για την Ιταλική ε, περίπτωση, πολλή ενέργεια λιμένων θα μπορούσε να μπει ε, στο σιδηροδρομικό δίκτυο για το μελλοντικό σχεδιασμό, για την περιβαλλοντική ποιότητα, όλα αυτά ε, θα βελτιωθούν. Και σίγουρα η εντολή που θα έχω στο μέλλον νομίζω θα είναι να επικεντρωθώ σε αυτές τις πτυχές. Κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να αναφέρω στην Επιτροπή σας και ελπίζω να είμαι σε θέση να ανανεώσω το ραντεβού αυτό για τον πέμπτο διάδρομο του βασικού δικτύου τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις τεκμηρωμένες απαντήσεις που μας δώσατε. Τώρα να περάσουμε στην επόμενη έκθεση, αυτή του Ζήλ Σαβαρή, για το σχέδιο τα υπερθυμών 22, Δρέσδη, Αθήνα, Βουδα, μάλλον Αθήνα, Σόφια, Βουδαπέστη, Βιέννη, Πράγα, Νιρεμβέργη, Δρέσδη. Θα σε παρακαλούσα να παραμένει για την παρουσίασή σου στο όριο του διλέπτου. Αλλιώ δεν θα έχουμε χρόνο για την υπόλοιπη μερική διάταξη. Ε, συνάδελφοι, σα χαιρετώ όλου. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είναι η τελευταία φορά γιατί η δική μου αποστολή ολοκληρώθηκε. Ιδίω επειδή εξελέγει στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Οπότε ε, παρέμεινα στη θέση αυτή δύο-τρία χρόνια και νομίζω ότι έφερα εις πέρα στα κοντά μου. Θα σας κάνω λοιπόν μια παρουσίαση για να έχετε κάποια νέα προοπτική και κάποια νέα στοιχεία για την πολιτική μεταφορών μας. Για τον διάδρομο, για το σχέδιο 22, το σχέδιο προτεραιότητας 22, θα το ξέρετε με 7 κρατη να διασχίζονται και 8 διασυνοριακές περιοχές και δύο περιοχές που είναι πολύ διαφορετικές στην ε, διαχείριση των δυτική, με Γερμανία Τσεχία και Αυστρία και την ανατολική περιοχή, η οποία τελικά είχε πολύ περισσότερε ανάγκε και εκεί απαιτήθηκε μόνιμο συντονισμό μεταξύ των τεσσάρων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου ζήτησε να προεδρεύσω και σε μια ομάδα επαφή, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώ και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών συμμετείχαν. Εκεί έγινε ένα είδος πειράματος ως προς την διακυβέρνηση, πολλαπλή, ε, επειδή υπήρχαν πολλά κράτη-μέλη, αλλά και προκειμένου να βρεθεί μία και μόνη φωνή κοινή σε επίπεδο Γενικής Διεθνής ε, Περιφερειών με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Οργανισμού για τις Διασυνοριακέ Μεταφορές. Να ευχαριστήσω το σύνολο όσων συμμετείχαν όλα αυτά τα χρόνια στην δημιουργία και την διεξαγωγή των συνεδριάσεων αυτή τη ομάδα, η οποία πραγματικά πέτυχε το στόχο της νομίζω. Ως προς τη μέθοδο, καταρχάς ε, εκπονήσαμε δύο σημαντικές μελέτες. Μία, μία μελέτη για την καλή γνώση των διάφορων γραμμών, ε, γραμμική λοιπόν περισσότερο, και μετά για την ενδεχόμενη κίνηση και επιβατών και εμπορευμάτων, ώστε να υπολογίσουμε καλύτερα τις μελλοντικές μας ε, επενδύσεις. Ξεκινήσαμε με ποσά πολύ ε, υψηλά, με δύο ηλεκτροκίνητες οδούς, 140 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ότι σε ορισμένα τμήματα που θα χρειαστούν μόνο για τα εμπορεύματα, για τα φορτία, θα πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς αν θέλουμε πραγματικά ε, να γίνει ε, αποτελεσματική και σύντομη σιδηροδρομική μεταφορά. Τώρα, στα δυτικά είχαμε δύο ουσιαστικά σημεία επαφή, Γερμανία, Αυστρία και Τσεχία που επικοινωνούσαν εναλλάξει μεταξύ του. Αυτό το τμήμα σήμερα έχει υλοποιηθεί βάσει προτύπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά. Όμω, όπω θα δείτε, ω προ την υλοποίηση, αυτό που προβλέπαμε και προστανόμασταν τελικά συνέβη. Δηλαδή είχαμε πολλέ δυσκολίε για να διαχειριστούμε τη γραμμή που βλέπετε εδώ με κόκκινο, η οποία ε, είναι πολλά εκατομμύρια από τι επενδύσει μα με χώρε που έχουν ε, δυσκολίε στην ε, δική του χρηματοδότηση. Ήταν πολύ πολυκύμαντη αυτή η κόκκινη γραμμή, ε, είχε πολλές φυσικές δυσκολίες και ανομαλίες και δεν ήταν επιθυμητές οι γραμμές, τις φυσικές γραμμές επιθυμητές τις ονομάζουν αυτοί οι δικοί των μεταφορών. Οι γραμμές ήταν πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν, ήταν ανατολικά, ανατολικά ε, κατεύθυνση, η Κωνσταντζα, Πράγα, Βιέννη λόγω χάρη, αυτή η γραμμή που τώρα ολοκληρώνεται με δύο διασυνοριακές περιοχές που ακόμη δεν έχουν εναρμονιστεί πλήρως μεταξύ δύο κρατών μελών, αλλά εγώ πήγα εκεί, είδα τα διασυνοριακά αυτά τμήματα και βλέπω ότι προχωρούν. Επίσης, δύο μεγάλες επιτυχίες αυτόν τον άξονα από την ε, Μπέλα μέχρι το σταθμό της ε, Βιέννης, διότι ξέρετε ότι εκεί μιλάμε για ένα πραγματικό σταθυροδρόμι, θα υπάρχει ένα τέλειο σταυροδρόμι βορρά-νότου και ανατολής δύσης, και αυτός ο υπέροχος εξοπλισμός παρόλα αυτά μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα ως προς την εξυπηρέτηση της Βόρειας Τσεχίας. Διότι έχουμε ηλεκτροκίνηση κατά 160 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά δεν υπάρχει, υπάρχει πολύ περισσότερη κίνηση. Θα υπάρχει λοιπόν ένα μεταβατικό καθεστώς εδώ και ίσως και επιβραδύνσεις στην ε, οδό αυτή, οι οποίες Παρ' όλα αυτά ε, έχουν συμπεριλάβει το υψηλότερο πρότυπο που διαθέτουμε. Υπάρχει όμως εκεί πολλή ελπίδα για το μέλλον ως προς την κίνηση. Και μετά έχουμε και την περιοχή Βίλιμ Καλαθάτ. Τώρα προς τον Δούναβη που θα είναι εναλλακτικό τρόπος ως προς το δικό δίκτυο. Είμαστε μάλλον περισσότερο επιτυχεί για το ποδήλατο από ότι για τα συντροδομικά φορτία. Έχουμε δύο μεγάλα προβλήματα. Ω προ την πρόσβαση στι γέφυρε, θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα ερχόμενα χρόνια αυτό, γιατί οι συντροδρομικέ διασυνδέσει είναι πολύ αδύναμε. Τα κράτη-μέλη, ιδίω η Ρουμανία, έχει 8 ε, χιλιόμετρα πρόσβαση στον βορρά με 160 χιλιόμετρα την ώρα ω προ την κίνηση, αλλά με μέσο όρο 30 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή χρειάζεται κανείς ένα τετράωρο για 100 χιλιόμετρα. Λίγο παραπάνω από 100 χιλιόμετρα είναι τρομακτικό αυτό και σε ό,τι αφορά το βόρειο, την, νότια οδό της Βουλγαρίας με κόκκινο, η γραμμή αυτό, αυτή είναι ηλεκτροκινητημένη, αλλά με μία μόνο κατεύθυνση, οπότε πολύ αδύναμη. Για το Βίντιμ Καλαφάτ Μπορέτ, ε, Σα είπα ε, και πριν από δύο χρόνια ότι είναι ένα μεγάλο οδικό άξονα και για πολλά χρόνια θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν επιμείνουμε ω προ την πρόσβαση στη γέφυρα αυτή μεταξύ Ρουμανία, Βουλγαρία, η οποία δεν ε, δεν είναι άδικο αυτό θα έλεγα, δίνει περισσότερη πρόσβαση στην βόρεια θάλασσα παρά προς την νότια θάλασσα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια, ένας αγώνας δρόμου μεταξύ Βουλγάρων και Ρουμάνων για να γίνει πόρτα εξ Ανατολών και του χρόνου θα πρέπει να ξαναδούμε αν θα γίνει μια σύραγγα στο Βόσφορο. Στο Βόσπορο για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και από την Τουρκία. Δεν ήταν αρχικά μέρο τη εντολή μα αυτό, αλλά είναι νέο στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να διαταράξει τα πράγματα στην περιοχή και το οποίο θα ήταν καλό να το λάβουμε υπόψη από τώρα. Όλα αυτά δεδομένων των αξώνων ε, δυτικά, από δυτικά προ ανατολικά και του network που έχουμε δημιουργήσει για τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων. Κατά τα άλλα, δούμε τις επενδύσεις για αυτή την κόκκινη περιοχή, είναι σημαντικά τα ποσά που θα χρειαστούν. Ο ρυθμός της κίνησης δεν είναι απλώς ένα θέμα του, τεχνικό, αλλά έχει και θέματα Σέγγεν, ε, τα οποία συμπεριλαμβάνονται. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις διασυνοριακές περιοχές, ασχέτως του επίπεδου των προτύπων. Θα πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε, ότι χρειάζονται και τεχνικές γνώσεις και ανανέωση των γραμμών, αλλά υπάρχουν και φραγμοί πολιτικοί. Εμπόδια πολιτικά τα οποία παραμένουν. Οι Έλληνες έκαναν τεράστια δουλειά. Δείτε ότι είναι σχεδόν όλο πράσινο η πρόσβαση προς τον Πειραιά προγραμματίζεται για τα ερχόμενα χρόνια. Μιλάμε για πρότυπα άξιο θαύμαστα, είναι αξιοσημείωτο το έργο τους. Απλώς υπάρχει ένα θεματάκι με το βουλγαρικό σύνορο. Η γραμμή είναι μια γραμμή που περνάει από ένα φαράγγι στα βουνά, οπότε ήταν πολύ δαπανηρό να οργανώσουμε εκεί μια οδό με πολλή κυκλοφορία. Πάντως ε, τα πρότυπα που ακολουθούμε είναι για την ώρα ε, στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θέλαμε να φτάσουμε τα 160, αλλά είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε τα 140 ακόμα και τα επόμενα χρόνια με δύο κατευθύνσεις. Η οδός των Βαλκανίων πάντως είναι προνομιούχος για τη χώρα αυτή, μάλλον προνομιακής θέσης για τη χώρα αυτή. Βλέπετε εδώ στο χάρτη, στο πάνω μέρος, τα τμήματα Ανατολή-Δύση πολύ περισσότερα πράσινα από ότι κόκκινα και μετά βλέπω ότι στο βορρά νότο υπάρχει πολύ περισσότερο κόκκινο από ότι πράσινο. Ε, ουσιαστικά ανακεφαλαίνεται αυτό που σα έλεγα. Αυτό χάρτη. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά ως προς την διακυβέρνηση όπως σας έλεγα. Σήμερα, ποια είναι τα προβλήματα που παραμένουν. Πολύ γρήγορα, να ναι, ναι, το ξέρω πριν να συντομεύσω. Μιλάμε για τα διασυνοριακά τμήματα, Εκεί μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα και πιο γρήγορα. Ο καθένα επενδύει από την πλευρά τώρα δεν είναι σαφέ που μπορούν αυτά να συνδυαστούν. Μεγάλε δυσκολίε μεταξύ Γερμανία και Τσεχία ιδίω. Η Τσεχία έχει κάνει τη δουλειά τη από την πλευρά τη. Θα ήθελε να υπάρξει διέξοδο εργασιακή προ τη Γερμανία και με συντροδρομικέ γραμμέ που ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όμω οι Γερμανοί έχουν προτεραιότητε βορανότου. Και το μόνο που δέχτηκαν το Ομοσπονδιακό δηλαδή κράτος, δέχτηκε να γίνει ε, μια μελέτη δυτικά της Πράγας να ανανεωθεί μετά το 2020. Όμως, οπότε δεν είναι μέσα στο άμεσο επενδυτικό πρόγραμμα της Γερμανίας και η γραμμή που πάει από τη Σαξονία προς τη Γερμανία. Όμως όλα αυτά αυτή τη στιγμή έχουν, ε, πέρασει, έχουν μείνει σε τέλμα για τους λόγους που έλεγε και ανέφερε ο Πατ Κόξ. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες επενδύσεις και επιπλέον θα πρέπει ίσω να το δούμε. Υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στου άξονε βορανότου. Όμω το Core Network τα επόμενα χρόνια και στις επόμενες, ε, στην επόμενη περίοδο θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο ροστό και το Αμβούργο, αν επιδεικνυθεί αυτή η γραμμή. Τώρα, τα μεγάλα ερωτήματα που θα τεθούν στο μέλλον. Πρώτον, δεν νομίζω ότι πρέπει να ε, πάψει η μέθοδο διακυβέρνηση που βρήκαμε ω τώρα. Ε, διότι στην τελευταία συνεδρίαση τα ανατολικά κράτη-μέλη μου υπέβαλαν τα πιο ακριβή ε, επενδυτικά προγράμματα. Είναι κρίμα όλα αυτά να, ε, λόγω του κλίματος αβεβαιότητας να παραμένουν άχρηστα και ενώ έγινε τεράστια προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στόχευση των επενδύσεων αυτά να μην αξιοποιηθούν. Δεύτερο ζήτημα θα είναι η διακυβέρνηση των διαδρόμων των ίδιων, του συγκεκριμένου διαδρόμου. Προ, σταδιακά, εμείς οι ίδιοι τον ε, ΡΕΑ που διαχειρίζεται τον όγκο του φορτίων, τον συμπεριλάβαμε στι συζητήσει μα, αλλά μα είναι πολύ διαφορετική χρηματοδότηση από κάτω μέλο σε κάτω μέλο, με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό φορέα, τον ιδιωτικό τομέα σε κάποιε περιπτώσει. Οπότε το θέμα είναι πώ θα συνδυαστούν διαφορετικέ πολιτικέ μεταξύ των κάτω μελών. Ο συνδυασμό ε, τη ομάδα επαφή ε, PP22 με την κυβέρνηση του διαδρόμου που θα σχεδιαστεί στο μέλλον είναι κάτι που δεν είναι δεδομένο, αλλά καλό θα ήταν να υπάρξουν ε, πολλέ διασυνδέσει. Και μετά οι μεγάλε δυσκολίε. Ένα μεγάλο σχέδιο έχει ε, το μεγάλο αυτό σχέδιο μάλλον έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην ε, Βουδαπέστη. Στη Ρουμανία αυτή τη στιγμή φτάνουν τα πρότυπα. Από την Τσεχία έχει ξεκινήσει μεγάλος άξονας και στην, ε, στην Βουδαπέστη εντοπίζονται οι περισσότερες δυσκολίες. Ε, θα πρέπει να, να δούμε τι θα γίνει επίσης με τη γέφυρα Βιλικαλαθάτ, όπω σα έλεγα, με την ε, Βιέννη, με την ε, με το μελλοντικό συνδυασμό και τη διατροπικότητα μεταξύ σιδηροδρομικού δικτύου και Δούναβη. Ε, συνάδελφοι, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να είμαι αρκετά σύντομο όσο, όσο θέλατε. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σουάλοβο, πολύ στόμα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και έχω τις εξής ερωτήσεις. Περιγράφοντας τον άξονα αναφέρεστε σε μία ε, διαδρομή βορρά ε, Ανατολής Δύσης που είναι πιο πράσινη από τη βορράς Νότου. Ε, βέβαια όσο πιο πράσινος είναι ένας άξονας τόσο πιο έντονα φαίνονται τα κόκκινα εκείνα κομμάτια που δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και για το κομμάτι που αφορά τη Γερμανία και Τσεχία. Μεγάλο κομμάτι νομίζω του προγράμματος προτεραιότητων 22 ε, είναι και ο διάδρομος ε, Ρήνου Δούναβη. Εσείς λοιπόν στην εκθέση σας περιγράφετε τα γνωστά ήδη προβλήματα που αφορούν τις επενδυτικές προτεραιότητες διαφορετικές ε, μεταξύ ε, Τσεχίας και Γερμανίας και αναφέρεστε επίσης στην ανάγκη για μια πιο στενή και θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των διαφορών αυτών πλευρών. Αυτό το οποίο υπενήσεστε δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι μια πιο πολιτική, για να το πω ευγενικά, προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι εννοείτε τι θα βλέπατε, τι θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο και αν βλέπετε περιθώρια και βελτίωση στο, περιθώριο, στο, θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ρικέ, ο κύριος Ερτού. Ισμαήλ. Ευχαριστώ και ο Θεμεστομό. Δύο ερωτήσεις. Ευχαριστώ τα σας, καταρχάς κύριε Σαβαρή. Πρώτη ερώτηση. Είπατε ότι η διασύνδεση μεταξύ της και Γερμανίας, φαντάζομαι είναι Ρεμβέργης, Μάτρικ, Βερτσέκε, Χέπ δηλαδή, και Πίλσεν Πράγα, ε, δεν αποτελεί προτεραιότητα για τη Γερμανία. Ενδιαφέρον αυτό, ή μάλλον με ξαφνιάζει να το πω διαφορετικά, διότι στις διαπραγματεύσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές TNT, η γραμμή αυτή ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων και είχε δεσμευτεί η Γερμανία να προχωρήσει σε αυτόν τον άξονα. Ερωτώ λοιπόν, εάν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα δεσμευτικό σχεδιασμό μετά το 2020 και επίσης αυτό που αναφέρατε για το Βόσπορο, τη σύραγγα κατά το Βόσπορο, ε, σε αυτήν εμπλέκονται κονδύλια ευρωπαϊκά για την υλοποίηση. Φαντάζομαι ότι εννοείται την ε, σύραγγα Μαρμαράη. Έχουν λοιπόν διατεθεί ευρωπαϊκά κονδύλια και ανέποσα. Ναι, ευχαριστώ Κράμερ. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση και, και ευχαριστώ ιδιαίτερως για την φωτογραφία της γέφυρα στο Βιντέν. Είναι πολύ ωραίος ο ποδηλατόδρομος, καταπληκτικός. Ε, ως προς το δικό κομμάτι λίγο ακόμα λείπει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ ε, ευχάριστο ότι έχει προχωρήσει όσο και αν λείπουν κάποια σημεία ε, διασύνδεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα, διότι το κομμάτι της τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια από ελληνικής πλευράς έχει παγώσει σε Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης και για λόγους λιτότητας βεβαίως, γιατί τώρα πια είναι με τη λιτότητα μεγάλη πολυτέλεια ο, ο σιδηρόδρομος και γιατί να κάνουν ε, ε, ε, σιδηροδρομικές γραμμές οι Έλληνες με λεφτά ευρωπαϊκά τα οποία όμως έχουν παγώσει μεταξύ ίδιοι. Γι' αυτό λοιπόν και για να περάσω το θέμα της Πράγας θα ήθελα να ρωτήσω εάν η διασύνδεση Βιέννης αεροδρομίου και η συνέχεια της διαδρομής για την Βουδαπέστη, την Βρατισλάβα πρώτα και την Βουδαπέστη έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Γιατί από ό,τι ακούω δεν θα προβλέπετε ε, από τον κεντρικό σταθμό της Βιέννης μέχρι το αεροδρόμιο της πόλης ε, στην αεροδρομική διασύνδεση, ακόμη και όταν τελειώσει ολόκληρο το έργο. Υπάρχουν λοιπόν τέτοια προβλήματα ακόμα ή έχουν αντιμετωπιστεί. Νιρεμβέργη Πράγα για την ε, Γερμανία έχει τόσο μεγάλη σημασία που πάγωσε τα έργα η γερμανική εταιρεία. Προφανώ δηλαδή, μια διασύνδεση σιδηροδρομική, η οποία ήταν καταπληκτική, πρέπει να πω ότι προχωρούσαν τα τρένα με ταχύτερου ρυθμού από ό,τι σήμερα, θα καταργηθεί διότι η προτίμηση τίνει προ το ε, επιβατικό λεωφορείο, γιατί είναι ίσω πιο πολυτελέ, γιατί ίσω υπάρχουν άλλοι λόγοι το προτιμούν εν πάση Πάντως η Γερμανία δεν εκφράζει τέτοια βούληση για προώθηση αυτών των μέτρων. Έργα τα οποία προχωρούν και με πολύ μεγάλους, ε, με πολύ βραδείς ρυθμούς πρέπει να υλοποιηθούν. Ιδέλος δεν καταλαβαίνω τι είδους δεσμεύσεις είναι αυτές που έχει αναλάβει η Γερμανία για διαδρομές οι οποίες κοστίζουν τόσο όλα αυτά αλλά τελικά δεν υλοποιούνται. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν τι σας είπε ο Υπουργός. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Κύριο Σκούν, πρόεδρε ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαβαρίτο στον νηστή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανάλυση για την κατάσταση. Η βασική και κεντρική φιλοσοφία είναι οι άξονες ε, βορρά, νότου ανατολής, δύσης να συνδέονται και με τα κύρια λιμάνια και αυτό πιστεύω θα παίξει σημαντικό ρόλο το να κλείσουν δηλαδή κάποιοι ε, κενά, όπως σε παραδείγματι ε, από τη διασύνδεση στην, από την Αθήνα, την Κωνσταντζα, από την ε, Βουδαπέστη, από την Ιρεμβέργη Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίζουν. Τι, τι μοίρα θα έχουν, τι συνέχεια θα έχουν. Και αυτό βέβαια με τους άξονες από την Ιταλία μέχρι το Βερολίνο μέσω του Μπρένερ. Για τη Δρέσδη και το Βερολίνο ή τη Δρέσδη και τη Λιψία έχουμε ε, να κάνουμε με μια διαδρομή η οποία πρέπει καταρχάς να ανοίξει, να είναι ε, δυνατόν να, επιτραπεί η κυκλοφορία και με επίπεδο καλό, με υψηλή ταχύτητα, με ε, συνθήκες ασφαλείας. Νομίζω ότι έχουν προχωρήσει και πρέπει να κλείσουν τα κομματάκια αυτά του εις Βερολίνης ε, ε, Βερολίνου Δρέσδης, Βερολίνου Λειψίας. Αυτό λοιπόν θα μας πείτε τι υπάρχει εκεί πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε και πάλι το λόγο για την απάντηση. Συνάδελφοι, να μην σας ε, να μην σας απαντήσω ξεχωριστά, ε, να, να ομαδοποιήσω λίγο τι ερωτήσεις, γιατί πολλέ ήταν παρόμοιε. Για το θέμα των σχέσεων Γερμανίας-Τσεχίας, δίκιο έχετε κύριε Κούν, έγιναν πολλά έργα στη Γερμανία για την ανανέωση του δικτύου, μεταξύ Τρέζη Βερολίνου και στο τμήμα που πάει από το Βερολίνο προς Ανατολικά, την ίδια τη Γερμανία, αλλά το πρόβλημα που έχουμε σταθερά, επειδή ρωτήσατε πώς έπρεπε να αντιδράσουμε από πολιτική σκοπιά. Κατάφερα να αποσπάσω από το γερμανικό ομοσπονδιακό κράτος αποδοχή. Αποδοχή να, να εκπονηθεί μελέτη τοδοτούμενη από το κρατήριο της Αξονίας και την Τσεχία, ώστε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Άρα δεν μιλάμε για κλείσιμο ή πάυση, απλώς η Γερμανία είπε ότι δεν είναι άμεση προτεραιότητα και είναι άλλο πράγμα το αν υπάρχει διαφορά μεταξύ Τσεχία και Γερμανία για το τι δυναμικό θα έχει η γραμμή. Οι Γερμανοί λένε ότι έχουν, η τωρινή γραμμή έχει πολύ μεγάλη δυναμικό. Οι Τσέχοι λένε ότι έχει ήδη φτάσει σε κορεσμό η υπάρχουσα. Το Ομοσπονδιακό κράτο λοιπόν γνωρίζοντα ότι δεν ε, χρηματοδοτεί, επέτρεψε την επόμενη μελέτη, αλλά οι βασικοί χρηματοδότε είναι η Τσεχία και η Γερμανία με το κατοίκιο τη Αξονία. Απλώ οι πολιτικέ μου συστάσει. Από τη στιγμή που το αποσπάσαμε αυτό με διαπραγματεύσει σχεδόν διπλωματικού επίπεδου, τελικά βρισκόμαστε εδώ σε Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε διαγωνισμό για αυτή τη μελέτη. Και στον διαγωνισμό απορρίφθηκε η μελέτη. Μα περιπλέκει κάπω την ύπαρξη αυτό το πράγμα. Από εσωτερική σκοπιά. Έχουμε δηλαδή στην πράξη την, ε, την υποχρέωση να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία με διαφορετικά κράτη-μέλη, με διαφορετικές τοπικές κυβερνήσεις και εδώ όλο αυτό μεταφράζεται σε μια διαδικασία δημοσίας προμήθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναθέσω άμεσα τη μελέτη γιατί χρειάζεται να γίνει πρώτα διαχωνισμός με αν θέλουμε να το διορθώσουμε αυτό, πρέπει να είμαστε σε άμεσο διάλογο με την Γενική Διεύθυνση MOVE και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο σύντομη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μήνε και εξάμεινα για να συγκλίνουν οι απόψει και μετά να μην ε, παίρνει αρκά και όλη η προσπάθεια. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα και δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να απαντήσω. Πέραν αυτού, ε, κάτι για τον Νότο τώρα. Οι Γερμανοί δεν θέλουν τον Ιρεμπέργη Σέντινγκ να φτιαχτεί, γιατί το θεωρούν πολύ δαπανηρό. Θέλουν όμως να γίνει ένα μικρό τμήμα, Μάρκεβιτς Σέντικ, για να επισκευαστεί γραμμή που θα πήγαινε από το, από το Βορειολίνο προς τη Βαβαρία. Υπάρχουν λοιπόν μικρά βήματα πρόοδο από τη γερμανική πλευρά που συνάδουν με την πραγματικότητα, ε, προτεραιότητα για τις ε, μελλοντικές επενδύσεις, που δεν απαγορεύει και το να συνεχιστεί η όλη προσπάθεια μετά το 2020. Μια πρόοδο που θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και εμένα και η ΔΕ, ιδίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω να μην αφήσετε αυτήν την ε, ευκαιρία να εκμεταλλευτεί. Κάτι σημαντικό ακόμη για τους Γερμανούς ζήτησαν να φτάνει ο διαδρόμος αυτός και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις όχθες της Βόρειας Θάλασσης. Από το Ρόστοκ, από το Ροστόκ λοιπόν και το Αμβούργο θα υπάρχει ε, συνέχεια ως την Κωνσταντζα ουσιαστικά. Και ευτυχώς που οι Ρουμάνοι και οι Βουλγαροί έχουν κινητοποιηθεί. Έτσι υπάρχει μια καλή διάρθρωση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει σημαντική πρόοδος και αυτό θα εξυπηρετήσει και την Κεντρική Ασία. Οι Βούλγαροι μάλιστα έχουν ενσωματώσει πολύ καλά τις ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες και ε, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους ε, Ρουμάνους, με το Group 22, με την ομάδα 22 και το διασυνοριακό πλάνο προχώρα από την Ουγγαρία. Αυτό θα βοηθήσει και την, ε, το τμήμα των, της κίνησης στα σύνορα Τουρκίας-Βουλγαρίας. Κάτι μα ενδιαφέρει πολύ για το μέλλον. Για την Ελλάδα τώρα, έχετε δίκιο κύριε Γκράμερ, είναι το μεγαλύτερο ε, πρόβλημα, διότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά μια συνδρομική νήσο. Δεν δίνει πρόσβαση σχεδόν σε τίποτα στα βόρεια. Σας το είπα. Στη Βουλγαρία είναι μια γραμμή πάρα πολύ δύσκολη, ε, πολύ ορεινή και πρέπει να βάλουμε τόνους δυναμίτε για να φτάσουμε από εκεί προς την Βόρεια Ευρώπη. Για τα Σκόπια τώρα. Με την πολιτική γετνία σα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή, ακόμα και αν η γραμμή δεν ήταν τέλεια, χρειάστηκε περισσότερη εκδοδότηση από τη γραμμή ε, νότου-βορρά ε, που θέλαμε να πρωτοδοτήσουμε με, το, με την ομάδα 22. Αλλά ξέρετε, από την πλευρά τη Γεκοσλαβία, το πώ θα δείξουν τα σύνορα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν διπλωματικέ διατυπώσει για να δούμε πώ μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η βαλκανική γραμμή η κόκκινη γραμμή είναι πιο ε, μακρά σε χιλιόμετρα από ότι η γραμμή ε, την οποία αναφέρατε μέσω των Σκοπίων, όμω υπάρχουν όλα αυτά τα συνοριακά προβλήματα μεταξύ των κρατών μελών. Ε, θα δούμε πάντω πώ θα διαμορφωθεί και η διπλωματική γεωγραφία και η προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ό,τι φτάνει το, σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο τη Βιέννη και την πρόσβαση αυτό, δεν το έχω ακούσει καν να αναφέρεται. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κύριε Κράμερ. Ναι, αλλά... Από το Σίντινγκ δηλαδή συμφωνεί η Γερμανία να πάει στην Πράγα μέσω του Πίλσιν όμως, από βορρά αντί για νότο. Γιατί δεν μπορούν να εξηγιάνουν την ε, διαδρομή αυτή οι Τσέχοι. Ή τελικά εξηγιάνουν την άλλη διαδρομή που έπρεπε τους ή άλλους. Αυτή ήταν η εξήγηση αλλους αυτη ηταν η εξηγηση λεει Ο κύριος Σεβαρή έχει ε, ανακατασκευάσει το κομμάτι Πράγα-Πίλσεν σύνορο. Μεθόριος. Οι Γερμανοί συνενούν στα 15 πρώτα χιλιόμετρα μετά το Σέντινγκ για να φτάνει κανείς μέχρι το δίκτυο το γερμανικό αλλά για την ε, ανακατασκευή δεν θέλουν να φτάσουν μέχρι την Ιρεμβέργη. Άρα έχουμε 10-15 χιλιόμετρα από το Σέντινγκ που μας επιτρέπουν να έχουμε τους άξονες βορρά-νότου που έχουν και την προτεραιότητα για μας αλλά πάντως δεν θα γίνει ανανέωση, ανακαίνιση της γραμμής μέχρι την Ιρεμβέργη γιατί και κοστίζει και δεν είναι προτεραιότητα. Ε, δεν είναι προτεραιότητα η γραμμή βορρά-νότου, αλλά, ε, ανατολής δύση, αλλά βορρά-νότου. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σαβαρή. Ο συντονιστής έχει αγωνιστεί όπως όλοι οι συντονιστές μας ε, πολύ για αυτή την προσπάθεια, για αυτό το έργο. Όμως το πρόβλημα είναι ότι μας μένουν ακόμα εκθέσεις. Και κινδυνεύουμε να μην έχουμε αρκετό χρόνο για να τις κλείσουμε. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση και βέβαια καταλαβαίνω ένα θέμα πολύ περίπλοκο και δύσκολο να το εξαντλήσει κανεί, αλλά παρακαλώ όλα τα μέλη της Επιτροπής να δείξουν ε, προσοχή ώστε να μην εξαντλήσουμε το χρόνο. Τώρα, κύριε Σκλίσκα, για το έργο 27. Αγαπητέ Πάβελ, τελείτσικα, σε παρακαλώ, στο να το πει σύντομα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να κερδίσω έστω και χρόνο ή δυνατόν. Ξεκινώντας λέω ότι 8 και εδώ και 8 χρόνια εργάζομαι ως συντονιστής στο έργο αυτό. Και πρόσφατα αντελήφθη είναι ότι ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα. Έχω υποβάλει αιτήσια έκθεση, έχω παρουσιάσει αποτελέσματα, είτε που επιτύχαμε, είτε που θέλαμε να επιτύχουμε και δεν καταφέραμε. Πάντα, πάντως οι συζητήσεις μαζί σας ήταν χρήσιμες για μένα, με πολλούς τρόπους. Έχω δει αρκετές από τις πρωτοβουλίες σας. Την πολιτική διάσταση ήταν τί ιδιαίτερος και αλλά επιτρέψτε μου λοιπόν αυτά λίγα λόγια ε, θαυμασμού στην αρχή για να μην τα λησμονήσω στο τέλος. Θα ήθελα λοιπόν πολύ γρήγορα να περάσω στην ουσία των θεμάτων. Και την μέχρι τώρα περίοδο. Είχαμε ένα έργο χρηματοδοτούμενο βήμα το βήμα και αντίστοιχα και την πρόοδο βήμα το βήμα. Εξυγχρονίζουμε ακόμα γραμμή σιδηροδρομική με το ρωσικό σύστημα 15-20 mm στο πολωνικό λιθουανικό σύνορο Κάλμας με κάποιες δυσκολίες, αλλά λίγο πολύ μέσα στα χρονικά πλαίσια που είχαμε ορίσει με βάση τα αποτελέσματα μπορώ να διαπιστώσω. Η Εστονία έχει ολοκληρώσει εδώ και δύο χρόνια την ανακαίνιση. Η Λετωνία παρουσιάζει πρόοδο στα βόρεια και νότια της ε, πόλης της Ρήγα με καθυστερήσεις που γνωρίζετε ασφαλώς λόγω της ε, σοβαρής ε, ε, ύφεση στη Λετωνία, γενικότερα στην περιοχή, αλλά στη και για τη Λιθουανία έχουμε αυτή την, ε, αυτό το έργο που σας ανέφερα. Βλέπω λοιπόν ε, με αισιοδοξία ότι μπορούμε μέχρι τα τέλη του προσεχούς έτους να έχουμε ολοκληρώσει τους κύριους στόχους μας. Και αυτή είναι η θετική πλευρά της υπόθεσης. Ε, ολοκληρώνουμε όμως και τα θέματα σε πολιτικό επίπεδο, ε, το διάδρομο δηλαδή βόλτικα και το στόχο της ενσωμάτωσης της Βαλτικής που είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομικά ε, περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπόλοιπη εσωτερική αγορά ενοποίηση λοιπόν με υψηλής ταχύτητας ηλεκτροδοτούμενες σιδηροδρομικές γραμμές. Αυτή είναι η ευκαιρία που βλέπω εγώ. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος που διαβλέπω. Στόχος ο οποίος είναι αποδεκτός πιστεύω και τη χάνει υποστήριξη σε ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής. Αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι ο χρόνος εδώ έχει τεράστια σημασία. Και ιδιαίτερα να πω ότι πρόκειται για ένα παράθυρο ευκαιρίας ως προς την χρηματοδότηση με το νέο μέσον ε, συνδέοντας την Ευρώπη το 85% μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε μέσω αυτού, το υπόλοιπο 15% είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την ε, Τράπεζα ε, Επενδύσεων της Βορειάς Ευρώπης, των βορείων χωρών της Ευρώπης. Νομίζω ότι προβλήματα ιδιαίτερα με τις χώρες Βαλτικής δεν θα έχουμε. Μετά τις διαβουλεύσεις θα έχουμε μηδενικές πιστεύω συνέπειες ως προς την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των χρόνο αυτών. Η κατάσταση λοιπόν είναι πολύ θετική, επωφελής για κάθε πλευρά και τώρα θα πρέπει να περάσω στα έργα, αυτά που μένει να γίνουν και τα λιγότερο θετικά ή λιγότερο αισιόδοξα μηνύματα. Είμαστε σε μια φάση τώρα διαπραγμάτευση μεταξύ των βαλτικών κρατών της θέσπισης ενός, μιας σύμπραξης μίας δηλαδή ε, ενός νομικού προσώπου το οποίο θα υποβάλει τις αιτήσει για τη χρηματοδότηση επίπεδο Βαλτικής και για τον διάδρομο Βόρεια Θάλασσα Βαλτική για τη χρηματοδότηση. Το συζήτησαμε και την προηγούμενη φορά, έχετε δει πιστεύω και στην ετήσια έκθεση, τα μεγάλα πλεονεκτήματα της συνενετικής αυτής προσέγγισης και με δεδομένο το παράθυρο ευκαιρίας και το στρατηγικό στόχο που σας ανέφερα, ε, μου φαίνεται αποθαρρυντικό το γεγονός ότι στα κράτη αυτά υπάρχουν οντότητες, νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν καταβάλουν τον μέγιστο, τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια. Είναι μικρός ο κόσμος εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαθαίνω από διάφορους επιχειρησιακούς κύκλους ή άλλους ε, δηλώσεις του ενός ή του άλλου επικεφαλής ε, διοικητικού συμβουλίου αεροδρομικής εταιρείας ότι να εμείς θα θα κατασκευάσουμε μέχρι την, ε, το πολωνο σύνορο ότι όποιος πιστεύει ότι θα φτιάξουμε ευρωπαϊκών Πρωτεγραφών ε, σιδηροδρομική γραφή, ε, γραμμή μέχρι το πολωνολιθουανικό σύνορο είναι γελασμένος και αυτή είναι η ευγενική εκδήλωση της έκφρασης που χρησιμοποιήθηκε. Αλλά δεν πειράζει, α μην, μην είναι και ευγενής όποιο μιλάει για το θέμα αυτό, αλλά πάντω δεν δικαιούται να μιλάει κανείς ως ε, πρόεδρος μιας εταιρεία μονοπολί, κρατικού μονοπωλίου. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μονοπόλια, έχουμε με ιδιωτικοποιημένε εταιρείε και μπορώ να σα πω ξεκάθαρα τη γνώμη μου γιατί και εγώ από αυτές τις χώρες προέρχομαι και μου θυμίζει λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση τον παλιό καλό καιρό και που έχω ζήσει και στη δική μου την εποχή. Με καταπλήσει λοιπόν αυτό που βλέπω και ακούω. Τι συμβαίνει τώρα σε σχέση με τις συμφωνίες των εμπλεκομένων μετόχων και τις συμφωνίες που θα πρέπει να καθορίσουν την πορεία του σχεδιασμού και τις συνδρομικές γραμμές για τη Βαλτική. Οι τρεις χώρες λοιπόν της Βαλτικής που διαπραγματεύονται τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν παρουσιάσει πολύ, πολύ περιορισμένη πρόοδο και ίσως και αυτό να είναι και υπερβολή όπως σας το λέω. Πολύ περιορισμένη λοιπόν πρόοδος. Ε, κάθε απόφαση που έχει ληφθεί στη μία συνεδρία αμφισβητείται στην επόμενη συνεδρίαση. Και ίσως Κάποιες χώρες μεγαλύτερες, κάποιες, κάποιοι φορείς μάλλον στις χώρες αυτές μπορεί να έχουν πιο ισχυρό λόγο από την είναι την κυβέρνηση, το Υπουργείο το αρμόδιο. Από την άλλη όμως έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό έργο. Έργο το οποίο ναι ενσωματώνει τη Βαλτική αλλά χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό χρήμα και στόχο έχει να επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εμπορευμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την κάθε άκρη της μέχρι την κάθε άλλη άκρη της. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονεί κανεί για να μιλήσω ξεκάθαρα. Έχουμε επίσης εντοπίσει κάποια θέματα τα οποία ε, ίσως χρειαστούν σε διακυβερνητικό επίπεδο διαπραγματεύσεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά κάποια από τα θέματα θα χρειαστεί οπωσδήποτε να τα ενσωματώσουμε σε μια διακυβερνητική συμφωνία για την οποία και αρχίσει να γίνεται λόγος τώρα. Για μένα από εδώ και μπρος αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι μέχρι το τέλος του να υπάρχει συμφωνία. Εάν δεν τα καταφέρουμε, ε, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν θα είμαστε έτοιμοι για την προσεχή άνοιξη. Και την καμπάνα που θα χτυπήσει τότε. Ε, μέχρι το τέλος του χρόνου λοιπόν και ανεξάρτητος και της έκθεσης, της έκθεσης των όσων σας λέω σήμερα. Εγώ θα είμαι έτοιμος να σας ε, υποβάλω αξιολόγηση της προόδου και με τις δικές μου παρατηρήσεις, προσωπικές παρατηρήσεις, για το ποιος είναι υπεύθυνο ε, εφόσον δεν τηρηθούν τελικά οι στόχοι. Μπορεί να μιλάω κάπως πρόημα. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μα. Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση μέχρι τώρα δεν καταφέρνουμε νομίζω να τηρήσουμε του στόχου, να σεβαστούμε του στόχου. Και κλείνοντα κύριε Πρόεδρε, ξέροντα ότι έχετε πολύ περιορισμένο χρόνο, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονό ότι βλέπουμε κάποιε δυσκολίε που εμφανίζονται τελευταίο καιρό με συμφέροντα εδώ ιδιαίτερα, με θέματα που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ένα τελευταίο σημείο παραδείγματι είναι ότι ένα κράτος μέλος έχει φτάσει στις διαπραγματεύσει σε, διαπρα... διακυβερνητικό επίπεδο με το επιχείρημα ακόμη και της διασύνδεση της πρωτεύουσά του που δεν προβλέπεται καν στη γραμμή αυτή. Δηλαδή είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο το οποίο ανατρέπεται τώρα γιατί κάπως έρχεται και ανήκει θέματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Που είναι κομμάτι μιας νομοθετικής διαδικασίας που έχει περάσει μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένως, είναι σαφέ το, το τι μένει να γίνει. Η πρόοδο πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τα τέλη του 2013. Δεν βλέπω δεν το βλέπω πολύ πιθανό να επιτευχθεί ο στόχο, αλλά εάν χρειαστεί θα πρέπει να ε, ε, αποδώσουμε και τις σχετικές ευθύνες. Και, μια, ε, και αυτό που θα χρειαστεί θα είναι μια συμφωνία στέρεα, μια συμφωνία μεταξύ των εταίρων, ξεκάθαρη για να προχωρήσει το έργο. Τι τελευταίε εβδομάδε η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα κανθόδη, πρέπει να σα πω, με πολλέ πολιτικέ συζητήσει και εμπλοκές ε, και γι' αυτό και τα λόγια των ευχαριστειών και ε, η θετική εκτίμηση που εξέφρασαν νωρίτερα για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος Κάλλα γνωρίζει καλύτερα από ότι εγώ, ύστερα από 8 χρόνια, ε, το επιτελείο του, η Επιτροπή, οι αρμοδιότητε του έχουν διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ και είμαι έτοιμο να ακούσω και ερωτήσει Νομίζω ότι εκφράσατε διπλωματικά την δυσαρέσκειά σας, αλλά δεν είστε αποθαρρυμένος ακόμη. Ο κύριος Κράμερ, τον παρακαλώ όμως να περιστά δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Θα ήθελα να μου πείτε αυτή η εξυγίανση του κομματιού από το Τάλιν μέχρι το, τα σύνορα και μετά το Κόρνας. Θα είναι έτοιμη του χρόνου και με τι ρυθμού με τι ταχύτητα καλύτερα. Επίσης υπάρχει μια σιδηροδρομική, ένας σειρμός ο οποίος μπορεί, όπως συνέβαινε πριν από 50 ακόμα χρόνια, να διατρέξει ολόκληρο αυτό το κομμάτι της, ε, της διαδρομής ή θα πρέπει να γίνεται μεταπιβίβαση και μετα, μεταφορά. Για το κράονος τώρα. Η παλιά διασύνδεση, ξέρετε, περνούσε από τη Λευκορωσία και άρα έχει αλλάξει η διαδρομή, έχει τροποποιηθεί. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν έχω αυτό τον, αυτός ο χάρτης δεν είναι πολύ σαφής. Από το Λίστοκ περνάει στο Ελκ ή στο Κουβάλκι. Μέχρι το σύνορο. Σουβάλκι. Γιατί στο Ελκ ο Πολωνός Υπουργός υφυπουργό μου είχε πει ότι ναι, υπήρχαν κάποια θέματα για περιβαλλοντική προστασία, αλλά ήταν υφιστάμενη ήδη η διαδρομή, είχε ήδη χαραχθεί και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Ερωτώ λοιπόν εάν υπάρχει κάποια προόδος ή τελικά το 1,2 ε, δισεκατομμύρια που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Πολωνοί προτιμούν να το αξιοποιήσουν στα έργα οδοποιία γιατί δεν σκοπεύουν να κάνουν τίποτα για τον σιδηρόδρομο. Ερωτώ λοιπόν, έχει ξεκινήσει η γραμμή, έχουν αρχίσει τα έργα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα και αξιολόγηση του ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε μέχρι το Κάουνας, το γειτονικό Κάουνας. Και ξέρω ότι και η Λετωνία έχει πάρα πολύ σοβαρές αντιστάσεις εκφράσει για μια νέα, γιατί υπάρχει μια νέα γραμμή που ε, θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα ενδεχομένω για τους τουριστικούς προορισμούς της ε, ακτογραμμής και βέβαια και τα λιμάνια. Ε, αλλά αυτό έχει αξιολογηθεί και η, οικολογική, η οικονομική αξία που θα έχει τέτοια γραμμή όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για, τα, για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στο συντονιστή μας. σε ό,τι αφορά το Τάλιν και τα σύνορα. Όπως είπα, η γραμμή αυτή έχει ολοκληρωθεί. Εδώ και δύο χρόνια, λίγο πολύ μάλιστα. Δεν είναι βέβαια όπως έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιοχές, αλλού υπάρχει μόνο μία λωρίδα, Υπάρχουν ε, νησίδες όχι παντού, άλλοτε μπορεί να διασχίζεται από σιδηροδρομική γραμμή και η μέση της ταχύτητα είναι γύρω στα 100 την ώρα, λίγο πολύ. Μπορεί να κινηθεί και ταχύτερα βέβαια, αλλά τώρα σε ό,τι αφορά το σειρμό, α όχι, για το κάουνας, μέχρι τα σύνορα, έχει αναβαθμιστεί και δεν ήξερα κατά πόσον θα μπορέσουμε να έχουμε εξασφαλίσει αυτό το, την αναβάθμιση του εξοπλισμού. Πήρα διασφαλίσεις από τον Λιθουανό Πρωθυπουργό ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση, άρα δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ αυτό προς το παρόν. Για, τη... για το σειρμό τώρα δεν υπήρχαν τα τελευταία 20 χρόνια τρένα καθόλου, επιβατικά τρένα, για να απαντήσω τώρα τον κύριο Κράμερ. Μπορούμε, κύριε Κράμερ, να πάμε με ένα σύρμα πράγματι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό όμως. Το πρόβλημα είναι αν εφαρμόζεται πλήρως το σιδηροδρομικό πακέτο ή όχι. Δηλαδή, αν πραγματικά υπάρχει η απελευθέρωση. Και δεν μιλάμε μόνο για την περιοχή τη Βαλτική, αλλά και σε άλλε περιοχέ. Η νομοθεσία πρέπει να υλοποιηθεί. Και αυτό θα το δει η Κομισιόν. Έχω αμφιβολίες για το κατά πόσον έχουμε υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια, αλλά θεωρητικά ναι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Για το ΕΛΕΚ ή το εναλλακτικό πέρασμα. Δεν, είμαστε, δεν έχουμε μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα, γιατί τα προβλέπαμε όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, και στην πολωνική πλευρά του συνόρου με τη Λιθουανία, λόγω των ε, περιβαλλοντικών πτυχών που αναφέρατε. Έχει υποβληθεί μάλιστα μια μελέτη και ελήφθη απόφαση να περάσουμε από το ΕΟΚ. Άρα από περιβαλλοντική πλευρά αυτή η επιλογή είναι καλύτερη. Σημαίνει βέβαια και συμφωνώ μαζί σα ότι το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό, αλλά το να έχουμε στη διάθεσή μα ε, ε, έτοιμε όλε τι μελέτε μέχρι τα τέλη τη τρέχουσα δημοσιονομική περίοδου. Επίση, θα πρέπει να υπάρξει και προφορική δέσμευση των πολωνικών αρχών για το μικρό αυτό τμήμα μέσω του ε, ΕΛΚ, δηλαδή το τμήμα αυτό, το πολύ μικρό τμήμα, να ολοκληρωθεί εντό ε, τη αρχή του επόμενου, τη επόμενη επταετία. Τώρα για τη Λετωνία, ναι, πάντοτε αντιμετωπίσαμε και το είπα, θα το θυμάστε, ότι πάντοτε αντιμετωπίσαμε δυσκολίε με τι λετωνικέ αρχέ για την προτεραιότητα που θα έπρεπε να έχει ε, και ο Βορρασνότος και όχι μόνο Ανατολή Δύση που είναι για τι προτεραιότητε. Σήμερα, ε, θα σα το λέω, πριν από δύο εβδομάδε ήμουν σε μια συνάντηση όπου ήταν παρόντε οι πρωθυπουργοί των τριών χωρών από την Περδία του Λετονού και υπάρχει πολιτική δέσμευση και υπάρχει αυτό το σύμβολο για τη Ρήγα συγκεκριμένα, για την κοινοπραξία αυτή που θέλουμε, τη σύμπραξη να δημιουργήσουμε. Υπάρχουν ε, σίγουρα ε, κάποιες διαφωνίες, αλλά είναι θεμητά τα αιτήματα των ε, Λετωνών και οι διεκδικήσεις τους. Εγώ πάντως δεν βλέπω κάποια αντίσταση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει το σημείο της μη επιστροφής. Ε, τα προβλήματα δεν έρχονται άμεσα από τη Λετωνία πια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τελίτσκα. Ήταν ενδιαφέρον. Φαντάζομαι εσείς τα βλέπετε και επί το Ότι με το συνδεδρομικό πακέτο έχουμε κάποια θέματα. Κυρία Κάρλα Πέις τώρα θα πάρει το λόγο για να μας μιλήσει για τις πλωτές οδούς έτσι δροσιστούμε λιγάκι. Thank you very much, uh, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από το 2007 ως το 2013 επικεντρώθηκα σε δύο έργα. Και όχι από τα λίγο περίπλοκα. Πρώτα απ' όλα για τον ε, Μόζα τον Δανούβη, τον Δούναβη. Και τον Ρήνο. Εδώ χρειάζεται να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των ομάδων του περιβάλλοντος και όσων θέλουν να κάνουν κάτι για το Δούναβη. Κατά τα άλλα. Για τον Βόρειο Σικουάνα θα πρέπει να υπάρξει νέα στόχευση. Ελπίζω ότι σύντομα θα εκπονηθεί η σωστή μελέτη. Μετά λοιπόν από την μελέτη αυτή, ο Σικουάνας, ο Σεν του Βελγίου, τότε μπορεί να εξευρεθούν και κονδύλια και να βρούμε και χρόνο. Για τον... Για το Σένανορ λοιπόν θα τα αφήσουμε ως έχει για την ώρα για την διασύνδεση με τη Φλάνδρα και τη Βαλονία. Ξέρω ότι εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά γενικά είμαστε εντάξει. Για τη Φλάνδρα και την Ολλανδία υπήρξαν διπραγματεύσεις για το Τερνίζε, Αυτό λειτουργεί πολύ καλά και από τις δύο πλευρές και από τις δύο χώρες και θα είναι πανέτοιμο σε πολύ λίγο χρόνο. Τώρα για το Δούναβι. Πολύ περίπλοκος ποταμός, διότι είναι πολλές οι χώρες. Και κάθε χώρα ε, αλλάζει και κυβέρνηση και με το πέρας του χρόνου είναι πολύ δύσκολο να συζητήσει κανεί με μια χώρα αν δεν γνωρίζει τον Υπουργό. Που ο Υπουργό κάθε φορά είναι καινούριο. Τα πράγματα λοιπόν είναι περίπλοκα. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε κάθε φορά για να συναντήσουμε αμέσω έναν Υπουργό μόλι εκλεγεί, αλλά το αμέσω σημαίνει ένα τρίμηνο μετά την ανάληψη καθηκόντων. Οπότε πάντοτε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έγιναν κάθε είδου έρευνε, κάθε είδου προγραμματισμό, συζητήσεις, ό,τι μπορούσαμε το κάναμε ε, πριν τις περιβαλλοντικές μελέτες αδικτύπου, Οπότε νομίζω στην ερχόμενη περίοδο θα πρέπει επιτέλου να αναλάβουμε δράσει. Με τι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο, διότι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία το οποίο συναντούμε κάθε μέρα και είναι ένα εμπόδιο είναι η αποστράγγιση. Οι χώρες έχουν κάθε είδου πρόβλημα Και όταν προσπαθεί μια χώρα να ορθοποδήσει, είναι πολύ πιο δύσκολο σε χώρες να οργανωθεί με φέρει η ρημούλκηση που ε, πολλές φορές μπορεί να μην είναι απλή γιατί δεν υπάρχουν αρκετά σκάφη εδώ για την ε, ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρωθήκαμε περισσότερο στον εξοπλισμό, στα εργαλεία για το δημιουργήση που ίσως να είναι μια προτεραιότητα. Για την ερχόμενη περίοδο επίσης, οι πλωτές οδοί είναι πολύ σημαντικές, ειδικά να ακούσα τόσο είπε και ο κύριος Σαβαρή. Θα είναι ένα σύστημα μεταφορών που θα παίρνει όλο ένα και περισσότερη σημασία. Γιατί την περασμένη μόλις εβδομάδα επισκεφτήκαμε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και μα πήραν 4 ώρε 150 χιλιόμετρα. Τσούκου τσούκου πηγαίναμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ένα πράγμα σε αυτές τις χώρε. η ενίσχυση του δυναμικού τους. Ακούσατε από τον κύριο Σαβαρή τι συμβαίνει με το σύστημα με το σιδηροδρομικό σύστημα, το οποίο θα αργήσει να είναι έτοιμο, το δικό είναι εν μέρη έτοιμο. Το μόνο λοιπόν που μπορεί να είναι σύντομα έτοιμο είναι οι πλωτές οδοί. Ο δούναβη, Ο Δούναβης. Αν το πιάσετε από την περιβαλλοντική σκοπιά, είναι πολύ σημαντικό και έχουμε κάθε σεβασμό για τα περιβαλλοντικά ζητήματα μεν, αλλά είναι κάτι που γίνεται. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ σημαντικό να το θυμάμαστε αυτό. Τι γίνεται τώρα. Να ξεκινήσουμε με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στις αρχές. Η σχέση Βουλγαρίας-Ρουμανίας δεν ήταν κακή. Ήταν απλώς ανύπαρκτη. Τώρα νομίζω ότι κάτι καινούριο γεννάται. Το είδαμε από το 2012 περίπου. Και την περασμένη εβδομάδα, άλλωστε αυτό ήταν ο λόγος που επισκεφτήκαμε τις χώρες, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας και με Ρουμάνους υπουργού και με προλοντικούς φορείς Συντήθηκαν στη Σιλίστρα, στο Δούναβι και ήταν μια άριστη συνάντηση αυτή. Δήμαρχε και από τις δύο πλευρές. Πρώτη τέτοιου είδους ε, συνάντηση και οι πρωταγωνιστές του όλου έργου και όλοι είχαν κάποιο είδου ενθουσιασμό, κάποιο ζήλο για να γίνει επιτέλου κάτι. Τώρα κατάλαβαν ότι πρέπει επιτέλου να ε, αναλυθεί δράση προ όφελο των πόλεων και των πολιτών. Τώρα λοιπόν υπάρχει επιτέλου η αίσθηση που ξεκινά όχι από τις αρχές προς τι χώρε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις χώρες, αλλά επιτέλους από κάτω προς τα πάνω, από τον ίδιο τον κόσμο που ζητά να γίνει κάτι. Αυτό είναι μια πολύ καλή αρχή. Θα πρέπει να τρέξω πολύ για να προλάβω. Οι δήμαρχοι λοιπόν ενδιαφέρονται πολύ για την εδαφική ανάπτυξη. Με τα νέα εργαλεία που διατίθεται. Η συντήρηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το είπα ήδη. Είδαμε επί τρία καλοκαίρια η πλοήγηση να πάθει Τελείω στο τμήμα μεταξύ Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Ο Ρουμάνος Υπουργός ε, προσφέρθηκε μέχρι και να χρηματοδοτεί την ρήμονξη σε, σε αυτό το κομμάτι εφόσον χρειαστεί. Όμως θα πρέπει να υπάρξουν κοινά εγχειρήματα. Και ήταν επιτέλους η ώρα να το σκεφτούμε αυτό γιατί ο βιομηχανικός κλάδος χάνει χρόνο και χρήμα ελπίζει να υπάρξει μια πραγματική πλωτή οδό, όπου πραγματικά να υπάρχουν μεταφορέ. Τώρα θα συνοψίσω τα συμπεράσματά μου και τι συστάσει μου. Οι κατευθυντήριε γραμμέ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μιλούν για στενότερη συμπερίληψη των νέων διαδρομών στις διατροπικές μεταφορές. Εδώ είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε τις πλωτές οδούς, χρειαζόμαστε το Δούναβι. Η η διευκόλυνση διασυνδέοντα την Ευρώπη, το Connecting Europe και με το Horizon 2020 ε, αφήνει χώρο και για τον ιδιωτικό τομέα. Η περιφερειακή ανάπτυξη των ε, διαφορών επαρχιών είναι πολύ σημαντική. Αν και ήταν λυπηρέ τελευταίε πλημμύρε στο Δούναβι. Πλημμύρε οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί απλώ και μόνον αν υπήρχαν αντιπλημμυρικά μέτρα. Τι να κάνουμε τώρα για να λάβουμε μέτρα για τον Δούναβη. Θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα συνολικό ε, πρόγραμμα κάθε φορά. Πλοήγηση σε συνδυασμό με την άρδευση, την ε, ρημούλκηση και ούτω την μερικά μέτρα. Είναι σημαντικό αυτό για τους κατοίκους της περιοχής. Η συμμετοχή κρατών μη ευρωπαϊκή που εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική, με κατευθυντήριε γραμμέ που θα καθορίζουν μια κοινή προσέγγιση εφόσον υπάρχουν διασυνοριακά προβλήματα και όλα τα προβλήματα που έχει η Σερβία είναι πέραν των συνορών της, είναι πολύ τυχεροί Να το πω κιόλα αυτό. Είναι πρότυπο. Είναι πρότυπο γιατί στη Σερβία από την πρώτη κιόλα μέρα είχαν μη κυβερνητικέ και διακυβερνητικέ ομάδε, οι οποίε συζητούσαν όλοι μαζί. του συνεχάρει και ο WWF για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και έτσι θα συνεχίσουν ελπίζουμε. Θα υπάρξει μεταφορά από το πρόγραμμα RIF 2000, του Horizon 2020 μεταφορά κονδυλίων για να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που θα αυξήσουν την ε, οικονομική ελκυστικότητα των ε, πλωτών οδών. Θα πρέπει όλοι οι φορείς να εμπληκθούν σε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει όμως και ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η ανανέωση της συνθήκης του τη Σύμβαση του Βελιγραδίου για να ενισχυθεί και ο ρόλο τη Επιτροπή του Δούναβη και να αναλάβει ρόλο εδώ και δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαραίτητο αυτό, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν με του Ουκρανού. Το 2012 η δήλωση των Υπουργών στο Λουξεμβούργο στο τέλος του, στο, του καλοκαίρι του 2012 είναι πολύ σημαντική, πρέπει να ακολουθηθεί και θα την ε, επαναλάβουμε για να πάλι, λάβει πάλι επίσημο χαρακτήρα η σημασία της ε, συντήρησης και να δούμε τι θα γίνει ακριβώς με την ε, πλοήγηση ε, στο το επόμενο καλοκαίρι. Επίσης η επαναστόχευση του σχεδίου ΣΕΝ προχωρά, προχωρεί υπό την αιγύδα του κυρίου Παβό. Νομίζω θα σταματήσω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, για το... συνεχίστηκε η μελέτη. Απλώς η κυβέρνηση της Βαβαρίας και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισαν να επιλέξουν τη δρόμο Α την εναλλακτική μάλλον α, η οποία εγγυάται 200 ημέρες ετησίως σε ύψος ε, για 2,5 μέτρα ε, ύψος του νερού, στάθμης του νερού. Ε, εδώ να πούμε ότι και εμείς πληρώσαμε για την μελέτη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια εναλλακτική, θα, ποια μεταβλητή θα επιλεγεί. Απλώς θέλαμε να έχουμε πολλές μέρες και με τη στάθμη των 2,5 μέτρων. Θα υπάρξει κάποιο πόρισμα από την μελέτη, ελπίζουμε, και θα τα συζητήσουμε τα αποτελέσματα, προκειμένου να γίνει καλύτερη δυνατή χρήση της ε, μεταβλητής α. Ίσως να προσθέσουμε μέρες πλοήγησης, διότι η τεχνολογία προχωρά και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ε, ευφύς ιδέες από την επιστημονική κοινότητα. Για το κομμάτι που ανέφερε ο κ. Σαβαρή, θα μπορούσε να αλλάξει τελείως το σύστημα μεταφορών, τις ροές των μεταφορών στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Θα υπάρχουν δύο ροές, μία προς τα δυτικά και μία προς τη Ρωσία. Με τη νέα σύραγγα μπορεί να υπάρξει μετατόπιση των μέχρι τώρα στόχων μας. Και δύο λόγια, Πρόεδρε, για την Κωνσταντζα. Η Κωνσταντζα είναι ένας λιμένας με τεράστιο δυναμικό. Όμως, να πω και το εξής, ουδέποτε είδα λιμένα χωρίς ε, ε ξηρά πίσω του. Είτε υπάρχει πάρα πολύ κίνηση είτε οι πλωτές οδού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω λοιπόν που είναι το κομμάτι της ξηράς πίσω από την Κωνσταντζα. Αν θέλουμε να αναπτυχθεί η... τα λιμάνια της Βουλγαρίας και η Κωνσταντζα πρέπει κάτι να, να κάνουμε γι' αυτό. Κάτι να κάνουμε με τις πλωτές οδούς στη Ρουμανία. Αυτό είναι σημαντικό για τον κύριο Κράμερ, πριν μου θέσει όλες αυτές τις ερωτήσεις που αναμένω. Ναι, είναι η απάντηση. Και το θέμα είναι τι θα γίνει και με το γαλάτσι και τη διασύνδεση του με το Ρήνο. Εντάξει κύριε Κράμερ. Επειδή ξέρω τον κύριο Κράμερ, δεν νομίζω ότι γλιτώνουμε, θα θέσει ερωτήσεις. Ο κύριος Βαντάλεν και Κάντσιαν. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Όσο περισσότερο μπορείτε κύριε Βαντάλη. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πέις για τις προσπάθειές της. Έχω ένα ερώτηση για την πρόταση Σεν Σχέλντεν. Λέει ότι μάλλον θα έχουμε αίσιο πέρας. Ή το προαισθάνεστε απλά αυτό. Έχετε επιχειρήματα που το βασίζετε. Γιατί θα πάνε όλα καλά στο τέλος. Θα περιμένω να μου δώσετε την απάντηση. Δεύτερο, Το Νοέμβριο του 2012 έγινε μια ε, διάσκεψη, ήταν εκεί και η καγκελάριος Μέρκελ. Εκεί αναφέρθηκε ότι Ρήνος Δούναβης είναι προτεραιότητα για τη Γερμανία. Α, πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα. Η μελέτη μπλοκαρίστηκε, είπε η κυρία Πέις. Τώρα με την εναλλακτική, με τη μεταβλητή α, τι γίνεται κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχει σταματήσει η ναυσιπλοεία. Υπάρχει κάποια προοπτική ε, να έχουμε κυκλοφορία, να έχουμε κίνηση στο Δούναβι τι έγινε τελικά με αυτά που είπε η κυρία Μέρκελ, γίνονται πραγματικότητα. Ναι, όμω το θέμα δεν είναι ιστορικές προτάσεις στη Γερμανία, αλλά εν γέννη έχουν υποχωρήσει πολύ όπως και το κανάλι Ρήνου Δούναβη. Έχει ε, υλοποιηθεί μόνο ένα 10%. Εάν είχε υλοποιηθεί καλύτερα ένα 10% των προβλέψεων θα ήμασταν και ευχαριστημένοι. Πριν από 30 λεπτά πέρασα τον Δούναβη πριν από, ε, και έπρεπε κάθε 5 λεπτά να γυρνάω το καγιάκ μου έτσι ώστε να μην ε, συγκρουστώ με τα πλοία που κατεβαίνανε. Τώρα που ανέβηκα με το ποδήλατο στις όχθες του ποταμού ε, δύο ή τρία πλοία συνάντησα σε όλη τη διαδρομή, μια τεράστια διαδρομή που έκανα. Ο Δούναβης λοιπόν είναι πλωτός, είναι μεγάλο ποτάμι, έχει περιθώριο και χρειάζεται καλή διασύνδεση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οι ιστορικές πλωτές οδοί πάνε στον Ρήνο. Εκεί ακριβώς χρειάζεται να δώσουμε την έμφαση διότι είναι μεγάλο ποτάμι, φαρδί ποτάμι, βαθύ ποτάμι και για δε την Μέρκελ πριν από ένα χρόνο ήταν υπέρ ήταν υπέρ της ανάπτυξης της πρώτης οδού του Δουναβή, όπως και οι υπόλοιποι όλοι και στη Βαβαρία, ο Υπουργός και όλα αυτοί. Αλλά πρέπει να γίνει, να ληφθεί απόφαση εάν θα ε, καταστεί πολύ σύντομα πλωτός και για άλλου τύπου πλοία ο Δούναβης, αν θα πρέπει να περιμένουμε 20-30 χρόνια για να γίνει η ε, διεύρυνση. Για δε τις, ε, τους υδροφράκτες στο Βερολίνο, που είναι πολύ σημαντική και είχε πει και ο Υπουργό ότι είναι θέμα για το μέλλον και μας πηγαίνουν στο μέλλον και όλα αυτά. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ο σιδηρόδρομος από το Βερολίνο στη Βαρσοβία ε, οικοδομήθηκε κατά 180 χιλιόμετρα μόνο και τίποτε περισσότερο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές εσωτερικές πλωτές οδοί. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί και έντιμοι Μιλάμε για διευρωπαϊκά δίκτυα. Όταν ένα κράτος μέλος λέει όχι, πρέπει να είναι πεπισμένα, πρέπει να μπορεί να πείσει τα λοιπά κράτη-μέλη ότι έχει δίκιο και ότι είναι λογική η επιλογή του. Δεν μπορεί να λέει όχι και χωρίς άλλη συζήτηση να κλείνει το θέμα. Λοιπόν, η Γερμανία προκειμένου είπε όχι. Έστω, το δεχόμαστε όπως και ο κύριο Ερτού φαντάζομαι, αλλά να ξέρουμε και γιατί. Και ό,τι συνέπειες να υπάρξουν, εν πάση περιπτώσει. Κύριο Σερτού, Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριο Κράμερ. Με πρόλαβε ορισμένα πράγματα που θέλω να πω. Για την κυρία Πέτ, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Είναι η τέταρτη φορά νομίζω που σας βλέπουμε σε τέτοιου είδου συζητήσεις, τέταρτη φορά που υποχρεούμε να διατυπώσω δηλαδή, τις ίδιες ερωτήσεις και τις ίδιες παρακλήσεις. Μας δίνετε αυτά ωραία, μας δίνετε αυτά ωραία τεύχη με τις ζωγραφιές, με τους χάρτες, τους πολύχρωμους κτλ. Αλλά πλέον δεν μου φαίνεται πάρα πολύ αξιόπιστο και επί τη βάση των όσων γνωρίζω από το στράμπινγκ και όλα αυτά ότι πρέπει να κοιτάμε μόνο που λείπουν χρώματα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο τα διαφορετικά κομμάτια να τα παρουσιάζουμε στις πλωτές οδούς όχι με χρώμα απλώς, αλλά με αριθμό πόσα είναι τα πλοία τα οποία διασχίζουν, αξιοποιούν αυτές τις πλωτές οδούς. Το κόκκινο που βλέπουμε εδώ δείχνει ότι η Αυστρία, η Γερμανία δεν έχουν κάνει το κομμάτι που τους ε, αντιστοιχεί στις ευθύνες τους. Και πρέπει μεταξύ Στράουμπιν και Φερσόφεν να βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερες διαδρομές ε, από ότι σε άλλες περιοχές μπορεί να φαίνονται πράσινες. Ο κύριος Καντσάν, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την συντονίστρια Πέις για το έργο της. Κάποια στοιχεία ήδη αναφέρθηκαν. Εγώ πιστεύω πολύ στον προσανατολισμό των διευρωπαϊκών δικτύων προς τη μεγαλύτερη εντατικότερη συμμετοχή, αλλά θα πρέπει να γίνει και κάτι χειροπιαστό το σύστημα των πλωτών οδών, με περισσότερη συμμετοχή. Κοιτάζω και εγώ τους χάρτες αυτούς που μας ε, δώσατε κυρία Πέης αλλά δεν βλέπω τίποτε για τον ε, Πάδο. Ο χάρτης δεν καλύπτει το κομμάτι αυτό του Πάδου μέχρι το Μιλάνο. Ε, δεν είναι επικαιροποιημένο ο χάρτης αυτός, διότι διαβάζω, εντάχει το διάβασα, το φυλάδιο, αλλά υπάρχουν δύο-τρία κεφαλαιάκια αρκετά ασαφή. Τι γίνεται, έγινε κάτι στο μεταξύ, ή όπως την άλλη φορά να ελπίζουμε ότι μπορεί να φτάνετε ως το Μιλάνο. Η κυρία Σεναλόβα, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πέζ για την παρουσίασή της και να θέσω ένα ερώτημα για τις εσωτερικές πλοκές οδούς ε, στην Τσεχία, που ήταν και κομμάτι της εκθεσής σας. Εμείς δεν έχουμε πραγματικά πρόσβαση στη θάλασσα ως χώρα. Άρα τα σχέδια αυτά, τα έργα αυτά θα έχουν να κάνουν με την πρόσβαση μέσω του ποταμού Άλβα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυξανόμενη δραστηριότητα γύρω από τον Έλβα, το Δούναβι, βέβαια η νέα πολιτική εκπροσώπηση θεωρεί προτεραιότητα αυτό το έργο. Και επεξεργάζονται μελέτη σκοπιμότητας. Ε, εσείς πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο να γίνει αυτό το έργο. Σίλβια, δεν έχεις ακούσει, αλλά θέλεις να θέσεις ερώτηση, τέλος πάντων. Ναι, ευχαριστώ, Μπράιαν. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Πέις πώς βλέπει το νέο διάδρομο Ρήνου Δούναβη. Επίσης, τα έργα που είναι σε εξέλιξη σήμερα, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη βέβαια. Ποια είναι τα άκρο σημαντικά project για την ε, μεταφορά του ποταμού Δουνάβου. Η κυρία Πέις. εάν μου επιτρέπετε, να αρχίσω από το τέλος. Τα σημαντικότερα προγράμματα και κάτι που είπε ο κύριος Κράμερ, θα το απαντήσω ταυτόχρονα. Αν δείτε το Δούναβι, εγώ πάντοτε ξεκινάω από την Κωνσταντζα. Ξεκινάω από την Κωνσταντζα και βόρεια. Εάν η Γερμανία είπε όχι, και πιστεύει κανείς ότι είπε όχι στον Δούναβη, δεν ισχύει αυτό. Είναι τόσο μεγάλο το μήκος του Δούναβη στην ε, ε, Γερμανία, όσο και η απόσταση από, τον βόρειο, από τη Βόρεια Θάλασσα. Εάν λοιπόν την μπλόκαρε, μπλόκαρε την οδό αυτή, θα χρησιμοποιούσε και πάλι το δυναμικό ε, του Δούναβη. Το μεγαλύτερο κομμάτι του Δούναβη βρίσκεται εκτό Γερμανία και είναι 2.000 χιλιόμετρα που φτάνει στην Κωνσταντζα. Είναι πολύ σημαντικό για τι χώρε που βρίσκονται εκεί. Και κάποιες από αυτές είναι και ευερήκλειστες. Εάν δείτε λοιπόν τι κάνουν οι Σέρβοι ή το πόσο σημαντικό είναι για την Κροατία, ακόμη και οι παραπόταμοι είναι σημαντικοί και σε πολλούς επιτρέπεται η πρόσβαση στη θάλασσα μέσω του Δούναβη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία πραγματικά αυτή τη στιγμή επιτέλους ε, δίνουν τα χέρια για να συνεργαστούν και να προχωρήσουν, να εξελιχθεί η κατάσταση από κοινέ προσπάθειες. Αυτό νομίζω ότι θα διευκολύνει τα πράγματα και επιτέλους θα καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Εάν λοιπόν πάω από κάτω προς τα πάνω, ναι. Στην Ουγγαρία έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά με το Βίλσο θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και τώρα εάν οι Γερμανοί δεν θέλουν να βελτιωθούν τα πράγματα, θα δούμε. Όμω στη Βαβαρία όλοι παραπονούνται για τα φορτηγά. Οπότε ή μία ή η άλλη. Εάν θέλει κανεί τα φορτηγά να πάνε πάνω στο νερό, θα υπάρξει φοβερή ανακούφιση για του ε, κατοίκου τη περιοχή. Εγώ ω Υπουργό θυμάμαι ότι οι Βαβαροί θύμωσαν, θύμωναν πάρα πολύ με τα φορτηγά, γανακτούσαν για την τόση κίνηση. Δεν θα το ξεχάσω όσο ζω. Δεν μπορώ λοιπόν να φανταστώ ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν θέλουν ε, τα φορτηγά, τέλος πάντων ε, τα κοντέινερ να πηγαίνουν σε, σε σκάφη, δεν μπορεί, το χωράει ο νους μου. Τι λέτε? Ναι. Όμως, εάν με το σιδηρόδρομο προς την Κωνσταντζα, δεν είναι πολύ το δυναμικό. Αυτό λοιπόν που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η πλωτή οδός. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να χρησιμοποιηθεί τελικά. Κυρία Σεναλόβα, με ρωτήσατε για τη δημοκρατία της Τσεχίας και αν υπάρχει εκεί λίγη περισσότερη δραστηριοποίηση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω όμως, και αυτό το θέλει απελπισμένα η δημοκρατία της Τσεχίας, πρόσβαση στο Αμβούργο. Δεν θέλουν να είναι πλέον περίκλειστοι. Εάν αυτό δεν επιταχθεί, τότε θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Δούναβι και να λειτουργήσει αυτό το τμήμα. θα πρέπει να μπορούν κάτι να βάλουν κι αυτοί σε ένα σκάφος και να πάει μέσω Δούναβη. Εδώ μπορεί να γίνει μια σχετική προσπάθεια. Όμως, η δημοκρατία της Τσεχίας θέλει να χρησιμοποιήσει στο Αμβούργο ένα τμήμα του για μεταβίβαση, για μεταβίβαση μάλλον φορτίου, εμπορικών φορτίων. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστεί εδώ η Γερμανία. Δεν μπορώ όμω να φανταστώ να θέλει η Γερμανία να τους μπλοκάρει. Είναι μια φοβερά επικερδής οικονομική δραστηριότητα και πολύ σημαντική για την Τσεχία. Κύριε Καντζιάν, ο πάδο. είναι ένα πολλά υποσχόμενο εγχείρημα. Βεβαίω και είναι, γιατί περίμενε πότε να ολοκληρωθούν τα προγράμματα του Σένενορ και του Δούναβη. Δεν έχει γίνει ακόμα πλήρω πλωτό ο πάδο. Βέβαια οι προσπάθειά ω τώρα είναι ιδιαίτερα επιτυχής. Εάν τώρα θα φτάσουμε και στο Μιλάνο, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε αυτό εάν πραγματικά το θέλουν οι Ιταλοί. Περισσότερο είναι θέμα δικό σας παρά δικό μας όμως. Εάν θέλετε θα ακολουθήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, διότι όλη η περιοχή είναι πραγματικά υπερφορτωμένη με οχήματα και φορτηγά. Κύριε Έρτουχ, μιλάτε για τα σκάφη. Κύριε Έρτουχ, για τα σκάφη και το δυναμικό του στόλου Έχετε δίκιο ότι η διάλυση δεν είναι η μόνη τακτική, διότι σύντομα, αν με ρωτούσατε πόσα σκάφη έχουμε, θα σας έλεγα σύντομα πολύ λίγα. Κύριε Κράμερ, σας υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να γίνει ο Δούναβης όλος πλωτός. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, ότι θα ήταν κάτι καλό. Έχουμε καλές σχέσεις με τις πραγματικέ ομάδες. Μιλάμε με όλους, μιλάμε μαζί τους, έχουμε επανειλημμένω συζητήσεις και προσπαθούμε να ε, ακούσουμε τις ανησυχίες τους. Η Ουγγαρία χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Η Σερβία είναι εντάξει. Με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία προχωρούμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εκεί τη σχετική δουλειά. Εάν τώρα με ρωτάτε τι θα γίνει με το Δούναβι, να σας πω ότι σίγουρα κάποια στιγμή θα πλέουμε σε όλο το μήκος του Δούναβι. Να σας πω βεβαίως ότι αυτό που με προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη είναι ότι δεν θέλει βαβαρία σκάφη στο κομμάτι της του Δούναβι. Κύριε Κράμερ, κύριε Κράμερ, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Η εταιρεία χρειάζεται κάποιο όγκο τα σκάφη να έχουν κάποια χωρητικότητα σε τόνους προκειμένου να είναι επικερδής η δραστηριότητά της. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε σκάφη που να αρμόζουν στις ανάγκες στα πρότυπα, τις προδιγραφές του Δούναβη, αλλά και να έχει και την ανάλογη χωρητικότητα το κάθε σκάφος. Έτσι είναι οι Εάν δεν έχουν χρήμα, δεν υπάρχει και μέλλον. Κύριε Φαντάλεν, είπατε για το για τον Έσκι. Νομίζω την βασική ουσία του θέματος, αλλά ισχύουν και τα δύο. Συζητήσαμε με ανθρώπους του Σένενορ ε, στο Ρότερνταμ και συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που έχουν οι κατοχώρες για ε, την κυκλοφορία σε πλωτές οδούς. Τα πάντα. Νομίζω ότι θα τους διευκολύνει αυτό. Εάν τα θέλετε, να σας τα στείλω και γραπτός για να τους τα δώσετε. Πρέπει όμως να τους βοηθήσουμε να λάβουν τις ορθές αποφάσεις με λίγο κόστος και ε, απλές. Ώστε να εξεύρουν και τα κονδύλια του ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσε να τους στηρίξει. Δεν είμαι η κυβέρνηση, αλλά έχω ε, θετικές ενδείξεις. Για το Straven Vilsover νομίζω ότι το συζητήσαμε αρκετά. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Τα μέτρα ως τώρα δεν ήταν πολύ αποτελεσματικά, αλλά πιστεύουμε ότι θα γίνει πιο αξιόπιστο αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ κύριε. Και τώρα έχουμε του δρόμο τη θάλασσα ο κύριο Βαλέντι Ολιβέρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ στιγμή. Τα τελευταία ξεκινήσαμε 31 έργα. Κάποια έχουν ολοκληρωθεί, κάποια συνεχίζονται. Εν όλο, πάντως, ήταν συνολικά Συμμετοχή σε 170 εκατομμυρίων ευρώ με συνολική επένδυση άνω του 1 δις Τα προγράμματα, λοιπόν, τα έργα τα οποία έχουμε μπορούν να, χαρακτηριστούν, μπορούν να κατανεμηθούν σε δύο διαφορετικούς τύπους παραδοσιακά που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση μεταξύ δύο λιμένων όπου έχουμε αρκετή επιτυχία, πιστεύω, σημειώσει. Εγώ προσωπικώ επεσκέφθηνα ένα από αυτά. Καλς Κλώνα, Δίνια. όπου έχουν υλοποιηθεί όλα τα έργα, έχουν ενισχύσει η διασύνδεση αυτή έχει ενισχύσει την κυκλοφορία μεταξύ των κρατών και έχει μειώσει τις ε, οδικές μεταφορές μεταξύ Σουηδίας, Δανίας και Γερμανίας χάρη στη σύνδεση Καλσκρόνα Κτίνια. Και άλλα τέτοια είδους έργα όμως συνεχίζονται. Ένας άλλος τύπος έργων είναι αυτό που ονομάζουμε έργα ευρύτερων ωφελιών γενικότερα δηλαδή έργα, στα οποία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όσο δεθούν περισσότερων εμπλεκομένων, γιατί η συμμετοχή πιστεύω στα έργα είναι και η κύρια διαβεβαίωση ότι μπορούν τα αποτελέσματα να ε, καταστούν ορατά αμέσω. Σε αυτά λοιπόν τα έργα ευρύτερης ωφέλειας μπορούμε να δούμε συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ διαφόρων ειδών στοχεύσεων. Καταρχάς της ασφάλειας, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες μεταφορές, ιδιαίτερα στη θάλασσα, ασφάλεια στη θάλασσα, και αυτή έχει επιτευχθεί για ορισμένα από τα έργα. Θα σας αναφέρω δεκτικά ένα. Το Μοναλίζα, υπό τον συντονισμό της Σουηδίας, όπου ε, τα επιτεύγματα αφορούν είτε την ασφαλέστερη ε, διακίνηση των πλοίων, είτε μελέτες που ε, που εξασφαλίζουν ότι η ρημούλκηση δεν θα είναι πρόβλημα, γιατί βέβαια η ρημούλκηση δεν εμφανίζεται ζήτημα μόνο στα, στους ε, ποταμούς αλλά και στους λιμένες. Αυτά λοιπόν. Το θέμα ήταν της ασφάλειας καταρχάς, να είναι ασφαλή τα ταξίδια. Δεύτερη στόχευση για τον ίδιο το λιμένα, την αποτελεσματικότητα, την ε, απρόσκοπτη λειτουργία του, όπου ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα είναι ο αριθμός των λειτουργιών που υλοποιούνται σε Εδώ λοιπόν αναπτύχθηκαν άλλα ε, έργα που έχουν να κάνουν μια μόνο μονοθυριδική προσέγγιση και διασύνδεση και εδώ μιλούμε όχι μόνο για μονοθυριδική προσέγγιση για τις τις λιμενικές υπηρεσίες Φερρυπίν τελωνίο, φυτογείνα, ακτινοτροφικός έλεγχος ε, και όλα, κτηνιατρικός έλεγχος και όλα αυτά τα οποία ήδη έχουν γίνει, αλλά και το Most for Most ε, έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί υπό τον συντονισμό της διοίκησης του οργανισμού Λιμένους Βαλένσια με πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα συνεχίζουμε προσπαθώντας ε, να υλοποιήσουμε ένα δεύτερο έργο B2MOS ονομάζεται και το οποίο αφορά την διασύνδεση μεταξύ των λιμένων και των δύο πλευρών αυτών. Δηλαδή ο λιμένα είναι πολύ σημαντικό για την επικοινωνία του πλοίου με την ενδοχώρα και τώρα προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση προκειμένου να έχουμε μια βελτιωμένη προσέγγιση στην ε, ε, αλυσίδα της επιμελητίας όχι μόνο μονοτροπικά αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα όπου χρειάζεται δηλαδή. Είτε πρόκειται για πλοία στο λιμάνι είτε πρόκειται για την αδοχώρα. Επίσης ένας δεύτερος στόχος ήταν αυτός ε, που έχει να κάνει με τα καύσιμα και βέβαια τις περιβαλλοντικές συνθήκες που μας απασχολούν ιδιαίτερα. Πέντε διαφορετικοί τύποι αντιμετώπιση του προβλήματος υβρέθηκαν ε, αντί για το κοινό ναυτιλιακό πετρέλαιο, το ντίζελ, το οποίο όμως είναι πολύ ακριβό και μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολύ βραχαίες, βραχαίες αλλά όχι στις μεγαλύτερες. Δεύτερον, η χρήση των λεγόμενων Scrabble στο αμπάρι του πλοίου, που είναι ένα πολύ βαρύ μηχάνημα και άρα προξενεί ζητήματα ε, ισορροπίας. Άλλες προτάσεις αφορούν τη βελτίωση των ε, Scrabblers και Και επίσης, καθώς δεν είναι κάτι το δοκιμασμένο, είναι νέο υλικό αυτά οι σκράπελες και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα στην ε, οξύδωση του λόγω του θαλασσίου νερού. Άρα πρέπει και την ε, μορφή και την τοποθεσία και το υλικό αυτών των σκράβλους να μελετήσουμε. Μεθανόλοι επίσης είναι μια λύση. Με περιορισμούς όμως πάλι στην ποσότητα ή με τι άλλο. Και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, έχει ιδιαιτερότητες. Έχει αχ, χαρακτηριστεί αυτοελεγχόμενη περιοχή εκπομπών, Βαλτική Βόρεια Θάλασσα Μάχη. Και άρα τηρούνται τα όρια έτσι τη στόχευση 2.15 εκεί, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθεί κάποια ε, όρια λιγότερο ίσως ε, άκαμπτα, λιγότερο αυστηρά, αλλά πάντως ε, πάλι στην ίδια στόχευση τίνει. Άρα έχουμε ιδιαίτερη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου, ιδιαίτερα για τη Βαλτική, όπου έχει ήδη εντοπιστεί, έχει ήδη διατυπωθεί ο σχεδιασμός του ελιμενισμού ε, σε όλη αυτή την περιοχή. Και για άλλους λόγους όμως, γιατί η Βόρεια Αμερική και ο Καναδάς έχουν αποφασίσει να, να ανακηρύξουν την Ανατολική και Δυτική όχθη της Βόρειας Αμερικής ε, περιοχές χωρίς φυσικό ε, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Άρα θα πρέπει να συνδυάσουμε δύο διαφορετικούς τύπους περιφερειών, βόρειο, ε, βόρεια Ευρώπη αφενός, ε, περιοχή δολαρίου από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Προβλήματα προκύπτουν ασφαλώς. Διαρωτώμεθε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους ή μικτούς τύπους ε, ε, καυσίμου, αν είναι δυνατόν ε, μόνο με υγροποιημένο φυσικό αέριο να περάσει, να διασχίσει ένα πλοίο τον Ατλαντικό. Θα δούμε. Πρέπει να το μελετήσουμε. Το τέταρτο στοιχείο που προωθήσαμε ήταν αυτό της κατάρτισης. το Moss, το έργο το οποίο έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει, το θέλαμε να διευρυνθεί. Τρεις χώρες μου έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν πρόβλημα ως προς την ε, κατάρτιση στον, ε, στα ναυτικά επαγγέλματα. Ωστόσο, χρειάζεται η εξασφάλιση προσωπικού, ε, ανθρώπινου δυναμικού και στα ναυτιλιακά επαγγέλματα βέβαια, αλλά και στη μεταφορά και γενικά την επιμελητία των καυσίμων. Γι' αυτό ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην επιμόρφωση και θέλουμε και να γενικεύσουμε ένα δίκτυο, γενικοποιήσουμε ένα δίκτυο επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων εκπαιδευτικών ανά την Ευρώπη που θα προσφέρουν το ίδιο επίπεδο κατάρτιση και επιμόρφωση. Και πέμπτον, όταν έχουμε να κάνουμε με την σωρευμένη γνώση που διαθέτουμε, πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρώπη είναι η περιοχή εκείνη του κόσμου που διαθέτει την περισσότερη γνώση για, τις, για τα θαλάσσια επαγγέλματα, τις θαλάσσιες μεταφορές και πολλά άλλα. Και έτσι θέλουμε να αναπτύξουμε και να γενικεύσουμε ένα δίκτυο που θα ενθαρρύνει ε, την ανταλλαγή αυτή των γνώσεων, της εμπειρίας, λαμβανωμένων υπόψη βεβαίως και των γνώσεων που σωρεύονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά Ινστιτούτα με την πρακτική απλή, ε, αυτή γνώση που έχουν όσοι εργάζονται στα λιμάνια. Έχουμε επομένως φορείς, ε, αυτά τα 31 έργα τα οποία προχωρούν, προβλήματα έχουμε φυσικά. Ίσως το πιο σημαντικό να είναι η διάδοση των αποτελεσμάτων μας και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο προωθούμε ιδιαίτερα τις ε, ενδιάμεσες συναντήσεις, τις συναντήσεις δηλαδή μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων αυτών έργων, ώστε να γνωρίζονται καλύτερα, ώστε να εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στα διάφορα προγράμματα Και έτσι λαμβανομένων υπόψη των όσων έχουν επιτύχει τα διάφορα project μπορούμε να δώσουμε λύση και στο περιπλοκό ζήτημα της διάδοσης των στοιχείων. Μίλησα εγκάρσια για όλα τα θέματα που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια. Θα μου πείτε πού είναι τα ζητήματα. Ζήτημα λοιπόν ως προ τη συμμετοχή στα έργα, μελέτες. Εκεί το είναι το δυνατό μα σημείο, το ενδιαφέρον και η γνώση που προσέφεραν. Και οφείλω να πω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τόσο έχουν επιτύχει. Πρόεδρος, μπορείτε να τελειώνετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν διαδραματίσει κεφαλαιόδη ρόλο και εν τέλει θέλω να εκφράσω ευχαριστίες μου στα μέλη της υπηρεσίας που με μεγάλη επιμονή υποστηρίζουν τα έργα αυτά και το προσωπικό που είχα στη θέση μου και στο οποίο οφείλω ότι έχω καταφέρει. Σε ευχαριστώ. Έχω δύο μιλητέ, του οποίου θα παρακαλώ να είναι συντομότατοι. Μόνο μισή ώρα πίσω έχουμε μείνει το πρόγραμμα. Τσικάω και Γέλα Σέντερ, σύντομα παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Από τα προγράμματα που μας αναφέρατε, δεν υπάρχει έργο που να έχει σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα. Το ίδιο ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε, διοργανώθηκε διαγωνισμός για έργα και υπήρξαν δύο προτάσεις από τη Ρουμανία. Η μία για τη δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου προς την Βόρεια Θάλασσα. Το προς τη Μαύρη Θάλασσα και εδώ ε, το έργο αυτό δεν επελέγει παρόλο που ήταν ισότιμο με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί δεν ξεκινάει κάτι που να έχει πρόσβαση και να προβλέπει διάδρομο προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συντονιστή και να κάνω τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, πώς εκτιμάτε το εξής. Οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα πιο πολύ έχουν κεντρωθεί στη βελτίωση των υποδομών και όχι υπηρεσίε. Δεν στήριξαν τόσο τι υπηρεσίε. Μάρκο Πόλο το τότε πρόγραμμα. Δηλαδή έγινε έδωθη μεγαλύτερο βάρος στις υποδομές. Δεύτερον, σχέσεις με τρίτες χώρες, βόρειοαφρικανικές, ή πιο, πιο ανατολικά από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς λέτε να πάμε πιο μακριά. Υπάρχει θετική εμπειρία όμως, μπορούμε να αναφέρουμε. Τέλος. Με τα άειλα θέματα, εκπαίδευση, εράσμους είπατε κιόλας για, το, για τον ναύτες που τόσο τους χρειαζόμαστε τι εμπειρίες έχετε να μας μεταφέρετε και τι συστάσεις θα έχετε να μας δώσετε να υπάρχει κάποιο νοτερικό στοιχείο σε όλα αυτά. Mr. Valenti. Κύριος Βαλέντε. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα. Πήγα στη Μαύρη Θάλασσα και στην Κωνσταντζα και στο Μπουργκάς και στη Βάρνα και έχω δει την κατάσταση εκεί. Έχω δει πως έχει κατάσταση εκεί. Εξήγησα ότι θα πρέπει να διατυπωθούν ε, συγκεκριμένες προτάσεις, σωστές προτάσεις για να προχωρήσουμε με το έργο. Στις συναντήσεις μας είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, δυνατότητες, αλλά όλες παρουσιάζουν δυσκολίες. Αν με ρωτήσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες, θα σας έλεγα κάτι που το συζητήσαμε και στις συναντήσεις. Η ενδοχώρα στην Κωνσταντζα. Υπάρχει σιδηρόδρομος από το 19ο αιώνα, ή τέλο πάντων αντιαρχές του 20ου. Αν με ρωτήσετε ποια θα ήταν για μένα προτεραιότητα πέραν των 30 χιλιόμετρων από Κωνσταντζα μέχρι τον αυτοκινητόδρομο θα έλεγα ότι έπρεπε να λιανθεί και να λιπανθεί. Ε, we have to ε, a group for Πάντως πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υποβληθούν προτάσεις και να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει και για τον Μπουργκάς. Ένα μεγάλο κόλπο όπου δεν μπορούν να ελμένιστούν πολλά σκάφη μεν, Μάλλον θα μπορούσαν ε, θεωρητικά να είναι στον πολλά σκάφη, αλλά είναι πολύ δύσκολη η διασύνδεση με το υπόλοιπο της χώρας. Δυνατότητες λοιπόν υπάρχουν. Εάν θέλετε να σας πω ποιοι είναι οι περιορισμοί, υπάρχουν πολλοί βασικοί περιορισμοί. Ο ένας, ο βασικότερος, ονομάζεται Βρυξέλλες και ο άλλος σχέσεις με τις άλλες χώρες τις ε, παράκτης χώρες της, ε, του ευξήνου πόντου, της Μαύρης Σω Ίσως να υπάρξει δυνατότητα να επιτευχθεί κάποια πρόοδος, όμως θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που για την ώρα δεν βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και προκειμένου να μπορούμε και να τις συζητήσουμε. Για να υπάρξει επιτυχία στην πρόταση επιτυχής έκβαση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το θετικό βήμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κυρία Γιάλα. Θέσατε κάποιες ερωτήσεις και θα σας πω αυτά που έχω να πω σχετικά, να σας πω τι προσπαθούμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα η διασύνδεση με τις χώρες της Αφρικής. Πήγα στη Βαρκελόνη, μίλησα με την Ένωση της Μεσογείου και τους εκπροσώπους της και κοιτάξαμε τι θα μπορούσε να γίνει. Επισκέφτηκα το λιμάνι της Βαρκελόνης, της Βαλένθια, του Αλικάντε και τους ρώτησα τι διασύνδεση υπάρχει το ίδιο ισχύει και για τους λιμάνες της Ιταλίας. Από τη Γένοβα. Λόγου χάρη. Υπάρχει σύνδεση Γένοβα-Σαρδινία, Βόρειο Αφρική. Όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η μεταφορά γνώση, η, η ανταλλαγή γνώσεων υπέρ τη οποία τάσσομαι είναι πολύ σημαντική και για τα λιμάνια και για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν έχει να κάνει μόνο με τα της θάλασσας, ε, με τα επαγγέλματα των, ε, της θάλασσας, των ναυτικών. Περισσότερο έχει να κάνει με τη διοικητική διοργάνωση, με τους ανθρώπους που, είναι, που ζουν σε χώρες που είναι και λιμάνια και πρέπει και από τις δύο πλευρές, αλλά ιδίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουμε υψηλού επίπεδου επαγγελματισμό για να το επιτύχουμε. Σε ό,τι αφορά τις ε, υποδομές για το ΜΟΖ, έχουμε κάνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, όμως το παράδειγμα που σας έδωσα Το παράδειγμα αυτό είχε να κάνει με τις οδικές και συνδροδρομικές διασυνδέσεις με την υπόλοιπη χώρα το παράδειγμα Καλσκρόνα Γκδίνια. Και είχε μάλιστα να κάνει και με βελτίωση των σκαφών. Εάν λύσουμε το θέμα των διασυνδέσεων, οι αυτοκινητόδρομοι της θάλασσας θα λειτουργούν. Θα προτιμά ο κόσμος να χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί τις θαλάσσιες μεταφορές από ότι τις χερσαίες. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και την κυρία Πέης και τον κύριο Βαλέντε Τολιβέιρα για τις εκθέσεις σας. Και τώρα θα περάσω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως, την έκθεση, την γνωμοδότηση του κυρίου Καντσάν για το ΣΕΖΑΡ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα είμαι συνοπτικότατος διότι δεν θεώρησα ότι χρειάζεται να υποβληθεί τροπολογία για το κείμενο. Πρόκειται για μια απλή παράταση της ε, δραστηριοποίησης της εταιρείας Σέζαρ, του εγχειρήματο και προγράμματος Σέζαρ. Δημιουργήθηκαν και συγκεντρώθηκαν έτσι τα, τα απαραίτητα δεδομένα Ε, και μιλάμε για ένα εγχείρημα δημόσιο μια σύμπραξη κοινού δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, χρήσιμη για κάποια ερευνητικά προγράμματα που θα προ... για ακόμη 15 χρόνια και πολλές φορές για θέματα όπως ο έλεγχος της εναερίας κυκλοφορίας και προκειμένου η, η χορύπανση και η ατμοσφαιρική ρήπανση να περιοριστούν. Υπήρξε κεντρική διοργάνωση ώστε να υπάρξει συντονισμό και συνέπεια της επενδύσει και για τις χρυσέ υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες μάλλον εδάφου και για τις εναέριε υπηρεσίες. Εδώ θα πρέπει ένα μέρος του ΣΥΕΦ να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί και εδώ. Μιλώ τώρα για ένα ποσοστό γιατί ξέρουμε ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος δεν καταφέραμε να έχουμε μια ικανοποιητική λύση. Πιστεύω πολύ στο δυναμικό αυτών των, ε, στις δυνατότητες αυτών των παρεμβάσεων και στην αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Όλα αυτά για τους ε, υπεύθυνους της εναέρειας, κυκλοφορίας αλλά και για τα αεροδρόμια επιτρέπουν να γίνουν πολλές οικονομίες. Οπότε καλό θα ήταν να ακολουθηθεί αυτό το πρότυπο, να συνεχιστεί το πρόγραμμα για να επιτύχουμε τους στόχους του οποίους έχουμε θέσει. Ευχαριστώ Αντώνιο, ευχαριστώ που ήσουν σύντομο. Ε, το εκτιμώ. Κύριε Δανέλη, ε, ελπίζω να είστε σύντομοι συνάδελφοι. Το ξέρω θέλετε να πείτε αυτά που θέλετε, αλλά πρέπει να προλάβουμε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα ε, σε αυτά που είπε ο συνάδελφος Καντσάν. Συμφωνούμε απόλυτα. Το Σέζαρ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά μέχρι σήμερα. Ε, δεν συντρέχει λόγος να κάνουμε οποιαδήποτε τροποποίηση. Κάποια επιμέρους ζητήματα θα τα προτείνουμε ως τροπολογίες στην έκθεση για το ε, κοινό ευρωπαϊκό ουρανό που έρχεται ε, τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Thanks, Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ τη συντονίστριά μας και η συγκήτρια και ό,τι συγκήτρια για την έκθεση αυτή που δεν μπορούσε να έρθει στην ε, σημερινή συνεδρίαση. Ακούσαμε τον κύριο Καντσιάν. Όπως βλέπουμε εγκρίνει την πρόταση Κομισιόν, δεν καταθέτει τροπολογία. Συμφωνεί η συγκητριά μας και πιστεύει ότι το ΣΕΣΑΡ πρέπει να προοδεύσει και στα πλαίσια των νέων ουρανών. Έχουμε αυτά τα λειτουργικά μπλόκα, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ικανοποιητικά και γι' αυτό θα πρέπει να βοηθηθούν οι προμηθευτές στον τομέα των αερομεταφορών, θα πρέπει να συνεργαστούν. Γι' αυτό το ΣΕΣΑΡ θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να πρικοδοτηθεί με επαρκή κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να παραταθεί μέχρι το 2024 και να λάβει 600 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό αυτό και σωστός δρόμος, ολοκληρώνει με αυτή η συγκεντρία μα, είναι η υπερψήφιση πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Φώστε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία Να πω ότι στηρίζω απόλυτα αυτό που είπε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια. Σήμερα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που λέγεται Clearing the Air, ε, να καθαρίσουμε τον αέρα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα ανταγωνιστικό προς το ΣΕΖΑΡ πρόγραμμα και οι ε, US Airways κοιτάνε πώς θα μπορούσαν με αβιονική και με άλλο εξοπλισμό να εξοπλίσουν τα σκάφη για το επόμενο τζέμ, αυτό το ανταγωνιστικό προς το ΣΕΖΑΡ πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να φροντίσουμε να είναι όλα έτοιμα και είναι και ο κατάλληλη, κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο εισηγητής λοιπόν έχει την πλήρη υποστήριξη της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Baldwin από την Κομισιόν νομίζω λέγεστε. Μπορώ νομίζω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, κατ' εξαίρεση, και να ευχαριστήσω απλά ε, πολλάκις ε, τον εισηγητή και την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. 28 Νοεμβρίου λίγη προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας τη μεγάλη μέρα των ψηφοφοριών 17 Δεκεμβρίου. 28 Νοεμβρίου λοιπόν έχετε μέχρι τότε για να καταθέσετε τροπολογίες. Ευχαριστώ για το δεκπεραιώσαμε γρήγορα. Να έρθεις δύο τώρα είναι το επόμενο θέμα. Η ε, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πακέτο Ναγιάδες έχει να κάνει με δύο νομοθετήματα για παράταση της υπάρχουσας, της ισχύουσας νομοθεσίας και την ε, ανακοίνωση, τη σχετική ανακοίνωση νοιάδες που έχει να κάνει και με το σχετικό πρόγραμμα δράσης. Ως πακέτο είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε περισσότερο να επεξεργαστούμε καινοτόμες, βιώσιμες και αποτελεσματικές πλωτές οδούς και το σύστημά τους. Κάτι που είναι σημαντικό για πολλές χώρες. Είμαι Ολλανδή και ισχύει αυτό προφανώς και για τις κάτω χώρες. Θα καλωσορίσω εδώ την απόφαση των ε, συντονιστών για το πακέτο Ναϊάδες να διοργανωθεί ακρόαση στις αρχές Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, Μία παρατήρηση βάσει της πρώτης συνάντησης με τους σκιώδεις. Οι δύο αναθεωρήσεις αυτές που προτείνονται σε μεγάλο βαθμό είναι τεχνικού χαρακτήρα. Το πολιτικό περιεχόμενο έχει να κάνει με το πρόγραμμα δράσης Ναϊάδες, Το δεύτερο πρόγραμμα δράσης. Επειδή είμαστε σχεδόν στο τέλος της θητείας μας, είναι πολύ δύσκολο να ετοιμάσουμε και να προλάβουμε να συντάξουμε έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Διοργανώνουμε ωστόσο ακρόαση. Οπότε, σημαντικό θα ήταν να υπάρξει κάποια πολιτική καθοδήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των πορισμάτων της ακρόασης για το πρόγραμμα δράσης Ναγιάδες. Οπότε, θα ήταν καλό να υπάρξει ένα ψήφισμα που να προέρχεται από την Επιτροπή Μεταφορών και να υποβληθεί στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί, ώστε τουλάχιστον από πολιτική σκοπιά η φωνή μα να ακουστεί, να εκφράσουμε κάποια τοποθέτηση βάσει των όσων θα υποθούν στην ακρόαση. Διότι το να γίνει ακρόαση χωρί να υπάρξει κάποια συνέχεια δεν έχει και νόημα. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεν, αλλά όπως σε πολλού άλλου τομεί, έχει πάρα πολύ λόγια παρά δράση. Οπότε να δώσουμε την ισχυρή πολιτική στήριξη του Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Τροπή ώστε πραγματικά να δράσει. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει με ένα τέτοιο ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να συνοδευτεί και από τις δύο ε, αναθεωρήσεις. Ως προς τις δύο τώρα προτάσεις. Η πρώτη αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την δυνατότητα του στόλου. στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας υπήρξε ένα ε, ταμείο βάσει των παλαιών κανόνων, χρήματα τα οποία ο ίδιος ο τομέας έχει συνεισφέρει και ε, επεξηγείται ότι τα χρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για να υλοποιηθούν κοινοτικά μέτρα και προκειμένου να αποφευχθεί η ε, περιττή αύξηση του δυναμικού του στόλου σε περίπτωση στρέβλωσης στις αγορές, αλλά και να ενισχυθεί ο στόλος, ιδίως εφόσον υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες και ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτό το στήριξαν και οι εκπρόσωποι του δικτύου για τις ε, Πλατές μεταφορές. Ε, αυτό ισχύει από το 1999 και παρόλο που κάποια κατημέλη και οι ίδιοι εργαζόμενοι προσπάθησαν να βρουν στόχους προκειμένου τα κονδύλια αυτά, τα χρήματα αυτά να δαπανηθούν, δεν το επέτυχαν, οπότε τώρα θα γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν επιτέλους προτείνει να διευρυνθεί το πεδίο και για την εκπαίδευση όλων των μελών του πληρώματος και την δυνατότητα χρήσης ε, των κονδυλίων για ανανέωση των σκαφών ή για τεχνικά προγράμματα που μπορεί να έχουν σχέση και με το περιβάλλον. Αυτός είναι ένας τομέας που πραγματικά χρειάζεται χρήμα. Οπότε καλό θα ήταν να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια προς αυτό το στόχο. Ξέρουμε όμω όλοι ότι μιλάμε για έναν κλάδο με πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει, με μέτρα τα οποία ουσιαστικά είναι δαπανηρά. Οπότε, καλό θα ήταν να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο το ταμείο, αλλά να επιδιώξουμε και μόχλευση, συνδυασμό με άλλα ταμεία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν ε, ο Πρόεδρος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το δουν αυτό, να δούμε τι μπορεί να γίνει ε, για να αξιοποιηθούν και άλλα κονδύλια. Ε, μπορώ να έχω δύο ακόμα λεπτά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Το ξέρω ότι βιάζεστε, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η δεύτερη πρόταση αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τα σκάφη των εσωτερικών πλωτών Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετικά νομοθεσία, αλλά και η CCNI και η Επιτροπή του Δούναβη, η UNC και όλες αυτές οι επιτροπές συνήθως συγκεντρώνουν τους ίδιους ε, εμπειρογνώμονες και ειδικού που επεξεργάζονται διαφορετικά νομοθετήματα ή προτάσεις. Προσπαθούν λοιπόν να εναρμονίσουν τα πρότυπα μεταξύ τους, αλλά αποκλήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν από πολλές απόψεις. Αυτό προκαλεί ασάφεια και νομική ε, αβεβαιότητα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μετά από συμφωνία με τη CCNR προτείνει να συγκληθεί μια κοινή μεικτή επιτροπή όπου οι εμπειρογνώμονες που είναι υπευθύνοι για τα ίδια τεχνικά πρότυπα θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εκπροσωπούν μάλλον ε, τις ίδιες απόψεις και στη CCNR και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε επιτέλους να υπάρξει σαφήνεια και να ισχύουν τα ίδια πρότυπα παντού. Αυτό θα ήταν μια πολύ σημαντική πρόοδος εφόσον ο στόχος είναι να υπάρξει συνεργασία μεταξύ CNR και των υπόλοιπων επιτροπών μακροπρόθεσμα της Επιτροπής του Δούναβη και των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, ώστε να μην υπάρχουν ε, περιττές ε, συγκρούσεις. Ε, σημαντικό λοιπόν είναι να στηρίξουμε αυτήν την προσέγγιση και μέσω νομοθεσίας ακριβώς με αυτήν την αναθεώρηση. Υπάρχει ένα παράρτημα στο κείμενο της αναθεώρησης που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές. Ως εισηγήτρια Κάπως ε, θα επιφυλασσόμουν να υποβληθούν τροπολογίες για το παράρτημα, διότι η εμπειρογνωμονε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων λέει ότι εκείνοι θα προτείνουν αναθεώρηση βάσει των τελευταίων στοιχείων, επιστημονικών στοιχείων, και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει μέσω κατακρισοδότησης πράξεων. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται και οδηγία για τον εξοπλισμό εκτός των οδικών και τα μηχανήματα μάλλον εκτός του οδικού δικτύου. Αυτό το περιμένουμε πολύ σύντομα για τα νέα μηχανήματα αλλά και για τις υπάρχουσες μηχανές. Θα επηρεαστεί όλο το σύστημα. Οπότε καλό θα ήταν να μην βιαστούμε. Ε, νομίζω για δύο τεχνικά ζητήματα ήταν μάλλον λίγο μακροσκελής η εισήγησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βορτμαν Κόλ. Παρακαλώ όσους θέλουν το λόγο να είναι σύντομοι. Έχω πρώτο τον κύριο Βαντάλη στον κατάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε την πρόταση. Πρέπει να πω ότι αισθανόμαστε μια μικρή απογοήτευση για τις ε, τεχνικές ε, προδιαγραφές παραδείγματι. Και απαιτήσει είναι 30 χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Και ακόμα δεν έχει κλείσει το θέμα τη κατανομή διότι το Νομίζω ότι θα μπορούσαμε πολύ πιο εύκολα να είχαμε καταλήξει μια λύση. Χωρί προβλήματα. Για το δυναμικό των στόλων, 35 εκατομμύρια ευρώ έχουν αφιερωθεί, κατά κύριο λόγο, έχουν, έχουν διατεθεί από τον τομέα. Νομίζω ότι πια πρέπει το Ταμείο να βρει μια εφαρμογή. Τα ποσά αυτά θα έπρεπε να επιτρέπουν στον τομέα να έχει σε θέση του μια αλφα για να κάνει τη δουλειά του. Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή εάν εάν υπάρχει πρόβλημα κατάρτισης ε, στον τομέα, ε, αρκεί αυτό σε αιτιολογία ή ως δικαιολογία για να αντληθούν κονδύλια που θα πάρει στην επιμόρφωση. Και πολύ καλά να γίνει. Χαίρομαι, με την κυρία, χαίρομαι τόσο μας λέει η κυρία Βότμαν Κόλ και συμφωνώ ε, ότι πρέπει να τοποθετηθούμε, να μπορούμε να τοποθετηθούμε και πολιτικά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τεχνικό πολύ το πρόγραμμα. Ε, πρέπει να διευρυνθούν αυτές οι προτάσεις εν του μέλλοντος και να προχωρήσουμε και μετά το ψήφισμα ε, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ερτού, εκ μέρους των Σελιστών και Δημοκρατών. Πολύ σύντομα παρακαλώ, διότι μου έχουν μείνει μόλις τέσσερα λεπτά και τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Πολύ σύντομα κι εγώ. Κυρία Βορτμαν Κόλ έχει Νομίζω ήδη δώσει κάποιε ενδείξει από την προηγούμενη εβδομάδα που συναντηθήκαμε. Πρόκειται για τεχνικέ προδιαγραφέ που πρέπει να εναρμονιστούν στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας. Εμείς στο εγγύς μέλλον σκοπεύουμε να κάνουμε μια ακρόαση, να ξανασυστήσουμε τα θέματα αυτά και εμάς σοσιαλιστές είναι πολύ σημαντικό το να προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό της εναρμόνισης, ήταν σημαντικό το θέμα αυτό και για μένα προσωπικά και ήθελα να διευκρινίσω προκαταβολικά ότι αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να ειστερούν σε τίποτα, ε, δεν μπορούν να προδικάσουν σε τίποτα τα, ε, όσα θα αποφασιστούν και θα κρυθούν στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο. για βάθος ποταμών και τα λοιπά. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πολλά θετικά πράγματα βλέπω να επιβεβαιώνονται πάντως και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ όμως και επιμένω ότι δεν πρέπει να προκαταβληθεί σε τίποτα ή να προδικαστεί σε τίποτα υπεραιτέρω συζήτηση που ήταν πολιτική. Ευχαριστώ, Ντεμπάκερ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Εκπροσωπώ την Γκεζίνε που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα. Η Γκεζίνε αλλά και όλη η ομάδα μα εν γέννη στηρίζει τι προτάσει αυτέ. Πιστεύουμε ότι μια κοινή δέσμη τεχνικών προδιαγραφών θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου θα την αυξήσει. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά το ταμείο, το αποθεματικό χρειάζεται ε, κάποια τροποποίηση. Ε, αν κανείς δεν μπορεί να εκπληρώνει τους όρους, δεν έχει νόημα για να λάβει αυτή τη βοήθεια. Συμφωνούμε με την ανάλυση ότι είναι τεράστιο το δυναμικό με τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Δεν το έχουμε εξοπλίσει ακόμη και πρέπει να το κάνουμε, όπως με το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη, το Connecting Europe. Η Γκεζίνη επίσης χαιρετίζει το γεγονός ότι το ταμείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε αυτά τα σκάφη να είναι πιο φιλοπεριβαλλοντικά. Θέλουμε να μειωθούν οι εκπομπές ε, καυσαερίων από τα πλοία και σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα αλλακτικά καύσιμα, πάλι έχουμε να βγούμε προς τα Δύο τεχνικές προτάσεις ε, είπατε ότι είναι ε, πρέπει να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της ε, εισηγητρίας για να βελτιωθούν τα κείμενα και θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη ιδέα για τις μελλοντικές προοπτικέ ε, προοπτικές των εσωτερικών της εσωτερικής ναυσιπλοίας. Εκπρόσωπος της Κομισιόν τώρα να είναι και αυτό σύντομος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος για μια φορά διότι νομίζω ότι τη στηρίζουμε απόλυτα την εισηγητριά σας, την κυρία Πόρτμαν Κόλ. Έκανε μια φανταστική σύνοψη των προτάσεών μας, ε, τα όρια του εγχειρήματος, τα περιέγραψε. Είναι ένα μετροπαθές εγχείρημα, μια μετροπαθές πρόταση προς τον κλάδο, αλλά σημαντική παρόλα αυτά, γιατί θέλουμε να διευκολύνουμε τη χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης. Σημειώνω το αίτημα και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να ταιριάξουμε καλύτερα αυτό το ταμείο με άλλες μορφές χρηματοδότησης, ερευνητική, χρηματοδότηση για έρευνα, που την ξέρουμε πολύ καλά, ή και άλλη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Connecting Europe. Σημειώνω επίσης την ιδέα να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των φορέων Υπάρχει ο μηχανισμός ε, ομοφωνία πράγματι, αλλά τελικά με συνένεση λαμβάνονται οι αποφάσεις. Διότι άπαξ και επιλεγεί μια ιδέα για να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του ταμείου αυτού, θα πρέπει όλος ο κλάδος να στηρίξει την ιδέα αυτή, γιατί όλοι συμβάλλουν με κονδύλια. Και οργανώσει πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές. Επομένως, θεωρώ ότι η τυπολατρική κατά κάποιο τρόπο διάσταση δεν είναι σημαντική του πώς λαμβάνονται αποφάσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δοθούν μεγαλύτερες δυνατότητες στον κλάδο. Φυσικά και θέλουμε να σας ε, βοηθήσουμε και με την ανακοίνωση να κάνουμε περισσότερα. Σίγουρα αντιμετωπίζει ο κλάδος δυσκολίες, είναι δύσκολη και η εν γέννη και ελπίζουμε στις συζητήσεις που θα έχουμε για την πρόταση αυτή να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και την ακρόαση αλλά και άλλες ε, δυνάμεις δυνατότητες που θα έχουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα από τεχνικής πλευράς απαντώ στον κύριο Ερτούκ σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τις τεχνικές προδιαγραφές. Αν δηλαδή θα έχουν να κάνουν και με το, τις διαστάσεις ε, του πλοίου, του σκάφου. Όχι αφορούν κάποια χαρακτηριστικά, αλλά όχι συγκεκριμένα τις ε, πλωτές οδούς, γιατί αυτό είναι αντικείμενο άλλων νομοθετημάτων. Thank you. I've got... Σας ευχαριστούμε. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 17 Δεκεμβρίου από την Κορίν. Η προθεσμία υποβολής των θα είναι 15 Ιανουαρίου. 2014 και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου. Όπως είπε η Κορίν, ακρόαση θα έχει διοργανωθεί στο ενδιάμεσο. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευτυχώς προλάβαμε. Τώρα θα αρχίσει η συνάντηση των συντονιστών.